Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei Καλημέρα σας. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση της επιτροπής μας. Η Πυρόεδρος, η κυρία Ματσόνη, ζητά συγγνώμη γιατί πρέπει να λείψει σήμερα το πρωί θα ήθελα να σας πω ότι μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Αυστριακού Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει αργότερα σε μία συνεδρίαση με την κυρία Ματσόνη και άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Σε σχέση με το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης προτείνουμε μία αλλαγή στο σημείο 15 σε ό,τι αφορά ε, την ε, η αναφορά 791 του 2008 θα αντικατασταθεί από μία συζήτηση τεχνική όπου θα συμμετέχουν ε, και τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στις 14-20 ε, Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι εγκρίνεται η τη διάταξη οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για τα σημεία 8 για την αναφορά 385 του 2011 σε ό,τι αφορά ε, την ε, αναφορά της κυρίας Μακμάνου, σημείο 13, αναφορά 1252-2011 σε ό,τι αφορά ε, την ε, τραγωδία αυτή σε ό,τι αφορά το σημείο 14 αναφορά 1347-2011 σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβαση στις πληροφορίες για τη σύλληψη και εκτέλεση του πατέρα ε, της κυρίας Γκόμε Ανκούλο κατά τον εμφύλιο πόλεμο τη Ισπανίας. Σημείο 16, αναφορά 1032-2010 σε σχέση με τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται οι μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων κατά την πρόσβασή του στα ισπανικά πανεπιστήμια. Ο κύριος ε, Μανουέλ Αλτεμίρ θα παρουσιάσει το σημείο αυτό. Κατόπιν, σημείο 17, αναφορά 1097-2011, η οποία αφορά τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος σε προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ε, Αναφέρον είναι ο κύριος Δεχάνα, σημείο 18 ό,τι αφορά τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μεγάλων ευρωπαίων υπηκών που προκύπτει από δίδακτρα που επιβάλλει ο Οργανισμός Γαλλικής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κυρία Κάρολιν Πέρσον θα εκπροσωπήσει τον αναφέροντα η οποία είναι βουλευτή στι Βρυξέλλε, σημείο 20, αναφορά 76-2012. Ο κύριο Όστιν δεν μπορεί να είναι παρόν, όμω έχει στείλει ένα γραπτό κείμενο που θα διαβαστεί στο όνομά του. Επίσης έχουμε και μία συζήτηση σε σχέση με την επίσκεψη ε, στην Ιταλία, τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία. Η συζήτηση αυτή θα λάβει χώρα πριν από τη συνεδρία των συντονιστών, πριν από τις 11.30. Τώρα, να περάσουμε στο σημείο 2 της ημερησής διάταξης. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων 12 Ιουλίου 2012 και 19-20 Σεπτεμβρίου 2012. Αν δεν υπάρχουν σχόλια. σε σχέση με το παραδεκτό των αιτήσεων. Έχει διανεμηθεί ένας κατάλογος σχετικός ε, πριν ε, από μία εβδομάδα και καθώς κανένα σχόλιο δεν εστάλει από τους βουλευτές, ε, θεωρούνται ότι εγκρίνονται και αυτές οι συστάσεις, ό,τι αφορά το σημείο 4 της ημερικής διάταξης. Αν κάποια μέλη θέλουν να αναφερθούν σε άλλα ζητήματα, παρακαλώ τώρα να είστε το λόγο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβληθεί κάποια σχετική πρόταση. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν τώρα στην μερσή διάταξη αυτή καθ' αυτή. Καταρχήν θα συζητήσουμε τη γνωμοδότηση σχετικά με τη βελτίωση των ωφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οικοδόμηση εμπιστοσύνη μέσω τη βελτίωση τη γνωστική βάση και τη ικανότητα ανταπόκριση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι η αρμόδια από τη ουσία Επιτροπή και η δική μα Επιτροπή έχει συντάξει μια γνωμοδότηση ο κύριος Τσίτσεστερ είναι ο εισηγητής. Καταρχήν να ζητήσω από τον εισηγητή να πάρει το λόγο αν το επιθυμεί. Παρακαλώ. Thank you ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαι έτσι τόσο γρήγορος όσο εσείς, αλλά θα προσπαθήσω να προτείνω στους σε αυτό το, το σχέδιο γνωμοδότησης. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια ισορροπία λοιπόν. Αλλά το σημαντικότερο ίσως είναι η παράγραφος 1 όπου βλέπουμε τον αριθμό των αναφορών ε, που αφορούν ε, περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτή είναι η εφετηρία μας προφανώς και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να στηρίξουμε τους αιτούντες όταν έχουν ε, τέτοιες ε, θεμητές ανησυχίες και όπως ε, ξέρουν οι συνάδελφοι όταν καλούμε τα κράτη-μέλη να είναι πιο ανοιχτά και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνεργασία υπονοούμε πως θα θέλαμε περισσότερη συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Τώρα, δεν ξέρω αν ε, μπορούμε να πούμε πως θα επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης οικονομίας και περιβάλλοντος. Εμείς θέλουμε πάντως οι κοινότητες τοπικές να έχουν λόγο όσον αφορά αυτή την ισορροπία καθώς αφορά την κοινότητά τους και το περιβάλλον τους και την άγρια ζωή. Και στο ίδιο πνεύμα λέμε πως θεωρούμε πως ε, οι πολίτες ε, που κατοικούν εκεί είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν καλύτερα τις ε, προτεραιότητες ε, της γειτονιάς τους και θέμε να ισχύσει στο μέτρο του δυνατού η αρχή της επικουρικότητας για περιβαλλοντικά ζητήματα. Μετά κοιτάμε την υπερφόρτωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ξέρω από την εμπειρία στον Ρωμανό Βασίλειο πως η τάση των εθνικών αρχών και των νομοθετικών αρχών και να είναι να προσθέτουν ε, διατάξεις ε, σε ευρωπαϊκά νομοθετήματα που μετά δεν είναι βεβαίως τόσο δημοφιλή και κατηγορούν, κατηγορούμε την Ευρώπη. Έχοντας κατά νου βεβαίως πως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί αντίσταση σε περιβαλλοντικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε θέλουμε τα κράτη-μέλη να μην ε, πηγαίνουν πέρα από τις απαιτήσει των οδηγιών όταν εφαρμόζουν ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Το σημείο 5 φαντάζομαι θα με ρωτήσετε γι' αυτό οπότε θα το προσπεράσω οπότε περνάω σημείο 6 υψηλά πρότυπα ενημέρωσης και διαφάνειας πρέπει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται και να, να βλέπει, να καταλαβαίνει το τι ζητάει η περιβαλλοντική νομοθεσία για να ε, υπάρχει και συνένεση των πολιτών για να εφαρμοστεί και η πολιτική. Καλωσορίζουμε τις ε, μελέτες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου, όμως ζητάμε να υπάρχει και πάλι, όπως είπα, αυτή η ισορροπία μεταξύ οικονομικών στόχων και περιβαλλοντικών στόχων. Και τέλος, προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους να συμμορφώσει καλύτερα την περιβαλλοντική, να συνδυάσει καλύτερα την περιβαλλοντική πολιτική με την κοινή αλληλευτική πολιτική και την κοινή γεωρική πολιτική. Οι καλύτερα αυτές οι δύο πολιτικές να συνδυαστούν καλύτερα με την περιβαλλοντική πολιτική μας για να ωφεληθούν ίσως κάποια ψάρια και η πανίδα και η χλωρίδα. Και τέλος, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το περιβάλλον με τρόπο απλό και φιλικό προς το χρήστη. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. με προς τους ε, φίλους μας που προτείνω εγώ να προτείνουμε στους φίλους μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τώρα κατά πώς θα δεχτούν είναι ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Τσίσσεστερ και τώρα καλώ την Επιτροπή να μας εκθέσει την άποψη ο Ζων Φρανσουά Ντεκλέτ από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο εισήγησης, συμφωνώ πλήρως με τα, την παράγραφο 1. Βεβαίως λαμβάνετε πάρα πολλές αναφορές, λαμβάνουμε πάρα πολλές καταγγελίες και γι' αυτό έχουμε τις ε, τρεις προτεραιότητες και την υλοποίησή τους που είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό που έβαλαμε στην ανακοίνωση του Μαρτίου είναι τρόποι για την διευκόλυνση της υλοποίησης από τα κράτη-μέλη. Πάρα πολύ συχνά ακούμε ότι το πρόβλημα είναι, το πρόβλημα των αναφερόντων είναι ότι προσπαθούν να βρουνε ε, μια λύση στο επίπεδο το κρατικό και τίποτα δεν υπάρχει διαθέσιμο. Γι' αυτό απευθύνονται σε εμά και σε εσά. Αυτό που προτείνουμε στην ανακοίνωσή μα είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε περισσότερε πληροφορίε ε, για του πολίτε να ξέρουν ε, τα δικαιώματά του ω προ την κατάσταση του περιβάλλοντο και να έχουμε περισσότερου μηχανισμού για απόκριση, για αντίδραση ε, αυτό είναι το θέμα της ανακοίνωσης, είναι ε, για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού νόμου. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται βεβαίως με το gold plating, την υπερφόρτωση με κανονιστικές υπερβολές. Ε, επίσης, μου η σχέση που κάνετε με το τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή ε, Περιφερειών επίσης ε, έχει μια εισήγηση και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε από την άποψη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και στην ανακοίνωση υπάρχουν μερικές ιδέες για εταιρικέ συμφωνίες, για εταιρικέ σχέσεις. Συμφωνούμε πλήρως λοιπόν με την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ δεδομένου ότι το κείμενο αυτό έχει αναλυθεί για πρώτη φορά εδώ, δίνω το συναδέλφους ε, ε, ε, που θέλουν να κάνουν σχόλια, κύριε Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη, είναι η Σαντρίν Μπελιέ, αλλά ε, είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτής της Επιτροπής. Δεν είμαστε μια παραδοσιακή Επιτροπή και γι' αυτό έχουμε πολλές απουσίες. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για τον κύριο Τσίτσεστερ. Θα έλεγα ότι συμφωνώ πλήρως για τρεις παραγράφους. Τέσσερις. Ένα, έξι, οκτώ και εννέα. Εξετάζοντας τις άλλες παραγράφους, ε, δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία ε, θα ήθελα βεβαίως να δω ε, την εισηγή σας, διότι όταν το διάβασα αυτό ε, θα πρέπει Greenpeace να έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν θα είχα αυτήν την πρόταση ότι θα είναι, πρέπει να είναι η Greenpeace που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Διαβάζοντας αυτά έχω την εντύπωση ότι, ότι αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται με ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό νόμο, αλλά σε τοπικό επίπεδο και αν αυτό αρμόζει στην τοπική κοινότητα, πολύ καλά με χαρά είδα την παράγραφο για την γεωργία και την αλία. Αλλά αν το αφήσουμε έτσι, αν ε, ο συντονισμός σημαίνει αυτό το πράγμα, τότε ξέρετε τι συμβαίνει. Έχουμε ε, μια μεγάλη συζήτηση στην Δανία, μια μεγάλη διαμάχη. Οι αγρότες ε, δεν ενδιαφέρονται αν κλείσουν ορισμένα πηγάδια νερού, αν η χώρα μου η ωραία γίνει μια έρημος διότι πιστεύουν ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα πώς να φροντίσουν, να μεριμνήσουν για τη φύση. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την άθλια κατάσταση στην Δανία σχετικά με τη φύση μας και τα τοπία μας. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα μας από αυτή την Επιτροπή στους αναφέροντες, δηλαδή να σοπάστε και να αφήσετε τους τοπικούς αλληλείς και αγρότες να ασχοληθούν με το θέμα. Ξέρετε ότι οι αναφέροντες έρχονται σε εμά θέλουν να έχουν ε, κάποια επιρροή ευρωπαϊκή ούτως ώστε να υπάρξει ένα υγιές περιβάλλον. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως ξέρω ότι είστε θετικός και κάνετε ό,τι μπορείτε για να υπάρχει κάποια ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όκεν, ο κύριος Ιάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα εκπροσωπήσω και την κυρία Κολάρσκα Μπομπένσκα της Χιώτης Γήτρια, η οποία επίσης δυστυχώς ε, απουσιάζει. Πρώτα απ' όλα επί της αρχής, ε, εγώ συμφωνώ με την έκθεση σε αντίθεση με την κυρία Άουκεν. Την ερμηνεύω και διαφορετικά. Εγώ για το σημείο 4 χάρηκα, όπου τονίζεται πως ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι σωστό να προχωράμε σε κανιστικές υπερβολές, γιατί έτσι υπάρχει ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν το αντιλαμβάνονται και οι πολίτες ότι συμβαίνει όταν στις δύο πλευρές των συνόρων ισχύουν διαφορετικά πράγματα Οπότε χρειαζόμαστε πράγματι ενιαία πρότυπα για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Θα μπορούσε επίσης να είναι και τίτλος «Εμπιστοσύνη μέσω περισσότερης πληροφόρησης». Και οι μισές αναφορές δεν θα έρχονταν καν εδώ πέρα εάν εφαρμόζονταν αυτός ο τίτλος. Γιατί έτσι είναι, αν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες δεν θα γινόταν πολλά πράγματα. και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ροή πληροφοριών και μεταξύ κρατών μελών και τοπικού επίπεδου. Εκεί που θα προτείνει αλλαγές η ομάδα μου είναι σε δύο πράγματα. Πρώτον, θα προσπαθούσαμε να βάλουμε την εξή πτυχή, δηλαδή αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να βελτιωθεί και μεταξύ των κρατών μελών, γιατί συχνά π.χ. μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας και από τις δύο πλευρές των συνόρων, έτσι. Ε, υπάρχουν κάποια αόρατα αλλά υφιστάμενα φράγματα στην ε, πληροφόρηση και πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ενημερώνονται αμοιβαία και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν έχει νόημα να αλληλογραφούν οι πρωτεύουσε. Οι πρωτεύουσε είναι πολύ πιο μακριά από το τοπικό επίπεδο. Και για τη ροή των πληροφοριών, όπως είπα, θα, εμείς θα, θα λέγαμε, γιατί πάντα αναρωτιόμαστε στην Επιτροπή όταν τοποθετείται η Κομισιόν Κομισιόν ε, εμείς κάνουμε ερωτήσεις, ε, ρωτάει η Κομισιόν τα κράτη-μέλη και έρχεται και μας απαντάει. Αλλά μετά έρχονται εδώ πέρα οι βουλευτές, οι επιτόποι και λένε «Μα ακούστε, εγώ αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα εκεί πέρα». Και ε, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση με κάτι άνεμο γεννήτρες έκανα ένα ερώτημα και έκανα την δοκιμή και καταλήξαμε στον άνθρωπο ο οποίος επεξεργάζεται το ζήτημα, ο οποίος δεν είχε ακούσει για ερώτημα της Κομισιόν. Οπότε ίσως το, ναι, το ερώτημα της Κομισιόν βέβαια πάει στο κράτος μέλος. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος μόνο για να απαντάει τις ερωτήσεις της Κομισιόν. δεν γίνεται έτσι. Πρέπει και η αρμόδια αρχή να, να εμπλακεί εκεί πέρα. Γιατί ε, έτσι εξηγείται μετά το ότι οι απαντήσει που λαμβάνουμε δεν είναι επαρκή. Οπότε θα πρέπει τα ερωτήματα αυτά να απευθύνονται στην υπηρεσία που μπορεί να απαντήσει. Όχι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνο για την αλληλογραφία με την Κομισιόν. και έχει έτοιμες απαντήσεις από το κομπιούτερ και τι στέλνει. Ε, ένα ερώτημα για το σημείο 5. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μετάφραση. Καταλαβαίνω το πρώτο μέρος που λέει τονίζει την επιτακτική ανάγκη κτλ. για ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων παραγωγή ενέργεια. Αναγνωρίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς επιπτώσει στο περιβάλλον. Αλλά μετά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Ζητάει από την αποκατάσταση του τοπίου μετά την ολοκλήρωση της ε, προτεραιότητας. Δεν ξέρω. Ε, μπορεί να είναι θέμα μετάφρασης. Γιατί σε γερμανικά δεν βγάζει νόημα. Αλλά κατά 99% είναι μια χαρά η έκθεση. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί όπως είπα πολλές ε, αναφορές φτάνουν εδώ πέρα γιατί δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό γιατί λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που συναντούμε καθημερινά στις δραστηριότητες της Επιτροπής μας, ε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Καταρχήν, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ανάγκη μιας κοινή ε, ερμηνείας όλων των υφιστάμενων κανόνων. Αυτό επιβάλλεται δεδομένου ε, του επίμαχου τρόπου με τον οποίο γίνονται οι ερμηνείες, όχι μόνο στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Επίσης, υπάρχουν αποκλίνουσες ερμηνείες μεταξύ κρατών μελών, όταν ε, πρόκειται για περιφελοντικά έργα διασυνοριακού χαρακτήρα. Λόγω των, ε, των περιβαλλοντικών αυτών προβλημάτων πρέπει να είναι και ομοιόμορφη η ερμηνεία. Η νέα οδηγία που ετοιμάζει η ΓΔ περιβάλλοντος θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιλαμβάνει αυτά τα πολύ απλά βασικά στοιχεία. Και θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό που να γίνεται αποδεκτός από όλα τα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια κοινή ερμηνεία όταν υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την προθεσμία απάντηση, την προθεσμία δράσης, ε, την προθεσμία υλοποίησης, θα πρέπει οι προθεσμίες αυτές να είναι ίδιες για όλα τα μέρη. Παραδείγματο χάρη, ένα παράδειγμα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο, το αεροδρόμιο τη Βιέννη. Όταν θα έχουμε επιλύσει αυτό το πρόβλημα θα έχουμε διασκεδάσει κάποιες αμφιβολίες που υπάρχουν, ότι δηλαδή κάποια κράτη και κάποιες περιφέρειες θα ήταν στόχοι της Επιτροπής Αναφορών. Σε ό,τι φέρουμε με το σχάρι, το σεβασμό της νομοθεσίας για την οικοδόμηση στην ακτή. Ε, θα έπρεπε να κάνουμε τα πάντα από το 2018 και από το 2014 με το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να πράξουμε έτσι ώστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσουμε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας, ε, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δούμε τι διδάγματα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Τσίτσεστερ για τη γνωμοδότηση που προετοίμασε. Η δική μας ομάδα επίσης θα καταθέσει τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η προσέγγιση και η φιλοσοφία της γνωμοδότησης μας φαίνεται πάρα πολύ λογική και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μποστινάρου. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Μπράκλεντ, αν έχει κάτι να προσθέσει. τότε να δώσω το λόγο στον κύριο Τσίτσεστερ για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν ε, και τους συναδέλφους για τα επικοδομητικά σχόλια. Πρέπει να παραδεκτώ ότι θα ανησυχούσαν η ε, κυρία Όκεν, ε, ήταν ικανοποιημένη με τα πάντα. Αλλά Ευχαριστώ την κυρία Όκεν για τα ευγενικά της λόγια. Παρ' όλα αυτά ελπίζω. Ε, μάλλον ε, έχει κάποια λανθασμένη εντύπωση. Εγώ δεν προσπαθώ να παρακάμψω την κοινωτική νομοθεσία. Αλλά θέλω να συνεισφέρω στο ότι θα νιώθουν οι τοπικές κοινότητες ότι έχουν ρόλο στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο ή στόχη. Ουσιαστικά δεν είπα κι εγώ ότι ήμουν ισορροπημένο. Θέλαμε μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των οικονομικών αναγκών. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο δυνάμει και της κατάσταση της οικονομική σήμερα. Ευχαριστώ τους αδελφούς για τα σχόλια. Μπορώ να πω ότι τα δικά σα σχόλια ήταν πιο ευπρόσδεκτα από τα της κυρίας Όκεν. κύριε Γιάρ. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε καλύτερα η πρότασή σας για τον τίτλο «Περισσότερη εμπιστοσύνη μέσω καλύτερης πληροφόρησης». Δεν μπορούμε όμως βέβαια τώρα να αλλάξουμε τον τίτλο. Νομίζω ότι τα όσα είπατε για την ανάγκη καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι κάτι σημαντικό και ελπίζω να παρουσιάσετε και μια σχετική τροπολογία που θα εμπλουτίσει το κείμενο. Τώρα η ερώτηση για την παράγραφο 5. Η παράγραφος 5 θέλει να μας υπενθυμίσει ότι χρειαζόμαστε πολλές πηγές ενέργειας και πρέπει να αναπτύξουμε νέες ικανότητες καθώς υπάρχει παροπλισμό σήμερα, γίνεται παροπλισμό σήμερα παλιών εργοστασίων, παλιών εγκαταστάσεων, ε, πυρηνικών, υδροελεκτρικών κτλ οι νέες δυνατότητες, οι νέες ικανότητες, το χάρη παραγωγή ολικής ενέργειας ή ε, ηλιακής ενέργειας, αλλά και πυρηνικής ενέργειας ε, και αερίου όπως χιστόλιθο, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Και αυτό που λέμε εμείς εδώ, τα κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να δώσουν προτεραιότητα στην αποκατάσταση του τοπίου μετά την ολοκλήρωση τη παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει. Ότι το τοπίο πρέπει να αποκατασταθεί στην κατάσταση που είχε πριν από την ανάπτυξη αυτή τη πηγή ενέργεια για την οποία μιλάμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ε, να ξαναγυρίσουμε στα πράσινα λιβάδια. Και ελπίζω ότι θα συμφωνήσει και η κυρία Όκεν με αυτό. Και ευχαριστώ τον κύριο Μποστινάρου για τι παρατηρήσει του για το ότι πρέπει να έχουμε κοινή ερμηνεία των κανόνων. Και εγώ θα καλωσορίσω για τις δικές σας παρατηρήσεις. Πρόεδρε, η κατάθεση των τροπολογιών ε, είναι στις 13 την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η προθεσμία. Έτσι λοιπόν, ανυπομονώ να λάβω τις τροπολογίες σας μόλις τις καταθέσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο κυρία Όκεν. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Νομίζω ότι όταν λέτε ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και στην οικονομία, αυτό εξαρτάται από το πόσο κοντόφθαλμος είστε στην οικονομία, πόσο βραχυπρόθεσμος. Έχω, βλέπω ε, πιο πακρόπνοα την οικονομία και τα παιδιά μου ε, και τα εγγόνια μου και τα παιδιά τους θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια υγιή οικονομία σε υγιές περιβάλλον. Αν έχετε λοιπόν μια τόσο κοντόφθαλμη οικονομία, οικονομική άποψη, πώς θα γίνει αυτό. Ο εισηγητής μας εδώ πέρα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία και η επόμενη γενιά έχει δικαίωμα και στα δύο, και στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Και το να, να τα επιτύχουμε και τα δύο είναι η ευθύνη μας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μπροστά στον κόσμο και όχι πίσω και πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό και δεν πρέπει να υπάρξουν αντιθέσεις. Γι' αυτό ακριβώ θεωρώ ισορροπημένη αυτή την έκθεση, γιατί δεν ρίχνει το βάρος σε ένα πράγμα, αλλά σε ένα πράγμα, αλλά προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα ενιαίο περιβαλλοντικό δίκαιο. Και αν, ε, όπως είπα, υπάρξει αγώνα για το περιβαλλοντικό δίκαιο, πρέπει να γίνεται στις στις Βρυξέλλες και όχι σε κάθε χώρα γιατί στη Γερμανία όταν έρχονται ε, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες εκγερμανίζονται δηλαδή τους φορτώνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και σας είπα τι, τι γίνεται στις μεθοριακές ε, περιοχές. Επικοινωνούν οι άνθρωποι και λένε «Μα τι γίνεται εδώ πέρα» Ευρώπη είμαστε, στη μία μεριά των συνόρων κάνουν το ένα και στην άλλη το άλλο. Και υποτίθεται ότι ισχύει το ίδιο δίκαιο. Να, έτσι χάνουμε αξιοπιστία. Γι' αυτό θεωρώ σωστή την έκθεση και ελπίζω. Να τα λάβει αυτά υπόψη της Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι σημαντική. Αν εφαρμοστούν τα πράγματα όπως αναφέρονται εδώ πέρα. Όπως είπα, θα γλιτώσουμε και πάρα πολλή δουλειά εδώ πέρα. Πάρα πολλές αναφορές δεν θα έρχονταν καν. Γιατί έρχονται γιατί ακριβώς δεν υπάρχει πληροφόρηση στα κράτη-μέλη. Θέλω να τη στηρίξω. Εγώ τη βρίσκω καλή την έκθεση. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τώρα που λέτε για κοντόφθαλμους. Καταρχήν εγώ είμαι ούτως ή ε, και αυτό είναι διακριτική μεταχείριση και αδικία. Αλλά τώρα για να σοβαρευτούμε λίγο. Έχω. Παιδιά ακόμα δεν, έχω, δεν μου έχει δώσει ο Θεός εγγόνια. Περιμένουμε με τη γυναίκα μου. Ε, περιμένουμε πολύ θεωρώ εγώ κατά την άποψή μου. Α, ντροπή σας, ντροπή σας. Λοιπόν, ε, για να μιλήσω σοβαρά, μα δεν έχετε μονοπόλιο στο ενδιαφέρον για το μέλλον ε, των παιδιών μας και των επόμενων γενεών. Όλοι μας, με τον τρόπο μας, ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ίσως έχουμε διαφορετικούς τρόπους, ε, απόψεις για το πώς θα, διασφαλίσουμε αυτό το μέλλον. Και ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε κάποια από αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. You know, not să Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία είναι 13 Νοεμβρίου για την κατάθεση των τροπολογιών και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Τώρα θα περάσουμε ε, στην ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Μεσελαβητή για την έρευνα σχετικά με την προσφυγή 2591 του 2010 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης. Ο εισηγητής είναι η κυρία Όκεν για το θέμα αυτό μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Αναφορών της Αυστρίας. Ε, κλήθηκε εδώ η κυρία Ούρσουλα Χάπνερ που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας, αλλά νομίζω ότι η αντιπροσωπεία θα έρθει λίγο αργότερα Γι' αυτό σας προτείνω να τους δώσουμε τον λόγο όταν φτάσουν. Τώρα δίνω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ούκεν. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα για την έκθεσή μου. Από όταν έγινε η πρώτη συζήτηση είχαμε κάποιες ε, συναντήσεις συνάντησα και εγώ κάποιους εκπροσώπους των Αυστριακών αρχών αλλά το θέμα εδώ πέρα δεν αφορά τις ε, αυστριακές αρχές αλλά τις σχέσεις μεταξύ Κομισιών και Διαμεσολαβητή. Τι συνέβη τώρα στην Αυστρία όταν ε, επεκτάθηκε το αεροδρόμιο της ε, Βιέννης δεν ε, προσπάθησαν να αξιολογήσουν ε, τις επιπτώσεις ε, παρά μόνο της πρώτης επέκτασης και θεωρώ πως είμαστε τώρα σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι αρχικά. Συναντηθήκαμε λοιπόν με την Κομισιόν και τον Μεσολαβητή και θα ήθελα να αναφέρω τα δύο σημεία στην έκθεσή μου που μπορείτε να τα δείτε αυτά. Είναι στο εκτιμώντας γιώτα όπου τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη εγκαίρως. Δηλαδή, εάν ξεχνάει κανείς ε, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα φτάσει μετά σε καταστάσεις δύσκολες και προσωπικά θεωρώ πως το όλο ζήτημα του να γίνεται μια αξιολόγηση ex είναι λανθασμένος ε, τρόπος ε, λειτουργίας και δράσης και, και η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να δώσει άδεια γιατί το, το εξπόστο εύκολα γίνεται post-mortem, μια νεκροψία δηλαδή. Ε, το άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά είναι το σημείο 10 και αφορά βεβαίως ε, την συνάντηση με τον Μεσολαβητή. Βεβαίως είναι συζητήσιμο το εάν ε, ισχύει νομικά το να πούμε πως ένα κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίσει ε, ανεξάρτητη μελέτη περιβαλλοντικών αντικτύπων το θέμα είναι πως ε, το Υπουργείο Μεταφορών στην Αυστρία έκανε και την αξιολόγηση και την επέκταση. Δηλαδή τον αξιολογεί κανείς τον εαυτό του δεν είναι και ότι πιο ανεξάρτητο. Οπότε αυτό το οποίο είπαν από πλευράς Κομισιόν είναι πως επαφίεται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες. Και εκεί πέρα υπάρχει μια γκρίζα ζώνη νομική, αλλά συνολικά στην νομοθεσία της Ένωσης υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Είναι στη χάρτα ορθής ε, διοίκησης ε, και τα λοιπά. Ένα από τα πράγματα, που αναφέρονται εκεί είναι πως ε, πρέπει κάποιος να είναι αμερόληπτος όταν κάνει αυτές τις αξιολογήσεις. και νομίζω πως ε, ήταν ζήτημα έλλειψης φαντασίας στην Αυστρία, ότι δεν σκέφτηκαν να ζητήσουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια μελέτη αντικτύπων για να δει εάν δηλαδή θα δεχόταν αυτά τα οποία έκανε το Υπουργείο Μεταφορών. Και εδώ πέρα είναι και η κριτική μου στην Κομισιόν και η Κομισιόν δεν το επεσήμανε. Και εγώ θα ζητήσω από την Αυστρία να έχει και λίγο περισσότερη φαντασία στο μέλλον. Για να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών. Οπότε υπάρχει αυτό το ζήτημα, το σημείο κριτικής. Υποστηρίζουμε επίσης και τον μεσολαβητή στην κριτική που ασκεί στην Κομισιόν και μετά τη συναντήση με την Κομισιόν έχουν αίσθηση πως τα πράγματα πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει λόγος να αποθαρρυνθούμε τώρα. Νομίζω πως ε, η Κομισιόν θα μας δώσει καλύτερα εργαλεία. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ δε στην ε, οδηγία για τις μελέτες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου μια πολύ σημαντική οδηγία και εκεί πέρα αναφέρεται και πρέπει να εφαρμοστεί το ζήτημα της ορθής είσαι έτσι ώστε οι πολίτες μας να θεωρούν ότι δεν τους ξεγελάμε στα περιβαλλοντικά χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια και η δυνατότητα νομικών μέσων. Και υπάρχει και η σύμβαση του άρχους για την εμπλοκή των πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Στο μέλλον ελπίζω να μην έχουμε αξιολογήσεις ex post ή τουλάχιστον να μην είναι όπως είπα νεκροψίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι συγχαίρω για την ε, εισήγηση, είναι ισορροπημένη για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν συμφωνούμε πλήρως με το σημείο 10 και νομίζω ότι η ουσία της συζήτησης, αν θυμάστε τι μας είπε ο Ομπουτσμαν εδώ στην Επιτροπή μας, ότι πρέπει η Επιτροπή να είναι πιο καινοτόμος, να έχει περισσότερη φαντασία. Και όπως εξηγείται στο σημείο 5, πιστεύουμε και πιστεύουμε ακόμα ότι ε, μπορέσαμε ε, να, ε, να συγχρονιστούμε με το χρόνο. Δεν, μπορέ μπορέσουν, ίσως πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα θέματα σχετικά με το conflict of interest. Βεβαίως μπορούμε ίσως να αναθεωρήσουμε την οδηγία για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, να έχουμε περισσότερα, ε, περισσότερες διατάξεις για την ρύθμιση των διαφορών, για συστήματα. Νομίζω εκεί και ελπίζω ότι με όλη ε, την εμπειρία που έχει αυτή η Επιτροπή ότι θα, περι, θα περιληφθούν όλα αυτά στην ε, ανάλυση για την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Όπως αναφέρεται στο σημείο 8 θα βελτιώσουμε τις εσωτερικές ε, μεθόδους εργασίας και ε, πώς να απαντήσουμε, να αντιδράσουμε στον Ombudsman. Έχουμε περισσότερη επικοινωνία με τον Ombudsman και με τους αναφέροντες. Ε, γι' αυτό ε, χαιρετίζουμε αυτήν την πολύ ισορροπημένη εισήγηση. Ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η έκθεση της κυρίας Όκεν. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή διατύπωση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο που μπορεί να χρησιμεύσει και για την περίπτωση αλλά και για άλλες ε, περιπτώσεις. Πιστεύω ότι το θέμα του αεροδρομίου ουσιαστικά μας έχει ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο και αυτό που συζητούμε στην πραγματικότητα είναι πώς να βελτιώσουμε τη λειτουργία και τις διοργανικές σχέσεις ε, μεταξύ της Κομισιόν και της δικής μας Επιτροπής Αναφορών και του διαμεσολαβητή. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα χρησιμεύσει το έγγραφο και για άλλες περιπτώσεις. Δεν... Ε, θα ήθελα να παραλείψω το ότι η κυρία και να αναφέρεται στις αυστριακές αρχές αμφισβητώντας ε, ε, τη φαντασία και η Κομισιόν αναφερθήκε επίσης σε αυτό το θέμα Ωραία. Νομίζω ότι σε αυτή την επιτροπή μπαίνουμε σε μεταφυσικά ζητήματα. Το ζήτημα της φαντασίας ε, δεν μπορεί να μετρηθεί. Ο καθένας μπορεί να το με διαφορετικό τρόπο. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι το ζήτημα της ερμηνείας. Και κυρίως ε, πώς ερμηνεύουμε την κακοδίκηση, τι είναι κακοδίκηση, κακοδιαχείριση και τι δεν είναι και επίσης το ποιος ερμηνεύει το αν πρόκειται για κακοδίκηση ή όχι. Και όπως προτείνει η κυρία Οκίνη, για να ξέρουμε αν υπάρχει κακοδιαχείριση ή όχι, θα πρέπει να προσφύγουμε σε ανεξάρτητους φορείς ή αν οι ίδιες οι αρχές κατά κάποιο τρόπο ή κατά κάποιον άλλο τρόπο έχουμε την εξουσία την αρμοδιότητα να ερμηνεύσουμε αν υπάρχει κακοδιαχείριση ή όχι. Είναι αλήθεια ότι ο ορισμός ε, της ε, κακής ε, της κακοδίκησης, της κακής διαχείρισης είναι κάτι αόριστο, δηλαδή δεν έχει οριστεί στα διάφορα έγγραφα που διαθέτουμε, γιατί δεν μπορεί να οριστεί. Προφανώς η κακοδίκηση υπόκειται πάντοτε σε διάφορες αποκλίνουσες ερμηνείες και κυρίως πρέπει να δούμε τι λένε τα θύματα αυτής της κακοδίκησης. Ίσως η συζήτηση που θα πρέπει να έχουμε είναι, είναι η εξή μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να ορίσουμε και να περιορίσουμε την έννοια της κακοδίκησης. Θα πρέπει να ορίσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται η κακοδίκηση σε κάθε περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι όση φαντασία και να έχουμε θα είναι αδύνατο να καλύψουμε όλες τις πτυχές μιας κυβερνητικής δράσης για να προσδιορίσουμε πότε υπάρχει κακοδίκηση και πότε όχι. Εγώ πιστεύω ότι όπως και να έχει η έκθεση, και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ την κυρία Όκεν. Η έκθεση λοιπόν είναι ισορροπημένη. Είναι μία έκθεση η οποία παράγει υλικό που θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στην περίπτωση αυτή αλλά και για τις διοργανικές σχέσεις μεταξύ θεσμών. Και κυρίω ε, θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να καθορίσουμε το ρόλο τη δική μα Επιτροπή. Και θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου γιατί η απάντηση που δίνει η Κομισιόν νομίζω ότι είναι μια λογική, μετρηπαθής απάντηση και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου. Μερικές φορές εγώ έχω ανησυχήσει και αισθάνθηκα και ντροπή μάλιστα όταν δημιουργήθηκε ένταση κάποιες φορές στην Επιτροπή μας και θεώρησα ότι δεν μας οδηγούσε πουθενά. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί όλα τα μέρη που παρεμβαίνουν, κυρίως η κυρία Ουκενική Κομισιόν, Νομίζω ότι τοποθετήθηκαν με τριοπαθώς και επιζητούν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εργασιών μας προκειμένου να ωφεληθούν και οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και να δηλώσω και την ικανοποίησή μου, γιατί νομίζω ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο και να δίνουμε και περιεχόμενο σε αυτή την Επιτροπή. γιατί θέλουμε να είναι αποτελεσματική. Έχετε το λόγο κύριε Μποστινάρου. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ο κύριος Μποστινάρου, αυτό που συζητήσαμε σήμερα δεν έχει να κάνει με τη στάση των Αυστριακών Αρχών, αλλά με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε ή έδρασε βάσει των υφιστάμενων κανόνων. Γιατί ο διαμεσολαβητής πρότεινε να εξετάσει εις βάθος το πώς υποχρεούται η Κομισιόν να εφαρμόσει τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες και συγκεκριμένα την οδηγία για την περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. είναι αλήθεια, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία λύση σου generis. Δηλαδή, περιβαλλοντική μελέτη δικτύπου ex post. Αυτή η λύση σου generis καλή είναι, αλλά από νομική σκοπιά δεν λειτουργεί. Γιατί ενώπιον οποιοδήποτε δικαστηρίου αυτή η λύση σου γκένερης ουσιαστικά αποτελεί κάτι που εφύβρατε και δεν υποχρεούνται οι δικαστές να δεχτούν μια τέτοια λύση. Θα έπρεπε λοιπόν να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να δρά πάντα βάσει των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται και που ισχύουν ενώπιον ενός δικαστηρίου γιατί τελικά θα πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες υπερβάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπογραμμίστηκε και από την εισηγήτρια την κυρία Ουκένη και από τους κοιόδης εισηγητές που συνεργάστηκαν στενά για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση για το θέμα αυτό. Και από τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Μαρτίνες υπόθηκε ότι η έκθεση αναφέρει και ορθώς τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν, να αποκατασταθούν με την νέα περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Καταρχήν, ο χρόνο απάντηση, ο χρόνο αντίδραση και από τι δύο πλευρέ, και τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Όπου οι διάφοροι πρωταγωνιστέ, διάφοροι φορεί ερμηνεύουν τι ε, ευθύνε του με ένα καινοτόμο τρόπο, με έναν εφάνταστο τρόπο που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα για τους πολίτες και τους αναφέροντες. Κατά την άποψή μου, η νέα οδηγία με επιτακτικό τρόπο θα πρέπει να θέτει προθεσμίες για να αναλαμβάνει δράση κομισιών και να απαντούν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, είναι επίση προφανές ότι ανέφερε ο μεσολαβητής ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ενώ εδώ είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τι είναι σύγκρουση συμφερόντων και αν ε, έγκυται αυτή η σύγκρουση συμφερόντων στην ε, αυστριακή νομοθεσία ή στην ευρωπαϊκή. Για να αποφύγουμε τις αμφισημίες και τη σύγχυση, η νέα οδηγία για την περιβολητική μελέτη αντικτύπου θα πρέπει με σαφήνεια να διευκρινίζει τι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Και επιτακτικά καλώ την Κομισιόν να σκεφτεί όχι μόνο ποιο είναι το καθήκον των ε, δημοσίων αρχών να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση, αλλά και των ιδιωτικών επενδυτών, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιώτες επενδυτές είναι αυτοί που υλοποιούν την περιβαλλοντική μελέτη δικτύπου και κατόπιν έρχονται σε εμά εντελώ ήρεμα και μα λένε ναι, έχουμε την περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου, αλλά πάρα πολλέ φορέ αυτή η μελέτη αντικτύπου σκόπιμα παρουσιάζεται ότι είναι ε, φιλική ε, απέναντι στον επενδυτή, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την ίδια την κοινότητα και για το περιβάλλον και υποχρέωση της νέας οδηγίας, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει υποχρέωση στη νέα οδηγία να διευκρινίζεται με σαφήνεια πώς η συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει να καθίσταται υποχρεωτική, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και έντιμη και συνεκτική. Διαφορετικά, ξέρω πολύ καλά από την εμπειρία της δικής μας χώρας. Ξέρω ότι από την επίσκεψη που είχαμε στη Βουλγαρία. Μερικές φορές οι αρχές, είτε οι κεντρικές αρχές είτε η τοπική αυτοδίκηση, βάζουν παραδείγματος χάρη μία έκκληση στο διαδίκτυο ε, για μια ακρόαση και έτσι παρουσιάζεται κατ' επίφαση η συμμετοχή των πολιτών και υπάρχει μια καλή οργάνωση, μια συνεδρίαση με, με διάφορους φίλους τους που παρουσιάζονται στην ακρόση και φυσικά η έκθεση θα είναι θετική. Αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον όλα αυτά τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν με νομικές διατάξεις όπου θα προβλέπω την υποχρέωση όλων των αρχών να σέβονται τους κανόνες και όχι να βρίσκουν λύσεις σου generis. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θέλω και πάλι να συγχαρώ την κυρία Όκεν για την εξαιρετική της ε, πρόταση. Ενώ δεν είναι εδώ. Α, εδώ είστε. Ευχαριστώ, Μάργαρετ. Και σχεδόν δεν χρειάζεται να βελτιωθεί η έκθεση με μη απαραίτητε τροπολογίε. Γιατί είναι πολύ καλή, είναι ουσιαστική, σοφή και προτείνει τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Γιατί η βασική αρχή του νόμου είναι ότι ο νόμος μπορεί να αναλάβει δράση για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου για τα ευγενικά σας λόγια. Παρακαλώ κύριο Σβέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως η συνεργασία με την εισηγήτρια ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία ως σκιώδης εισηγητής ε, Χάρηκα χθε που έλαβα το σχέδιο έκθεσης. Βεβαίω δεν μπόρεσα να το διαβάσω ακόμα αναλυτικά, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για μια ισορροπημένη παρουσίαση ε, των πραγμάτων που εμείς ε, μπορούμε να βγάλουμε ως συμπεράσματα από αυτή την περίπτωση ως Επιτροπή Αναφορών. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ στα επίπεδα στα οποία βασίζεται η ε, εργασία μας εμείς ευθύς εξ αρχής ε, είχαμε να κάνουμε με μια καταγγελία του μεσολαβητή κατά της Κομισιόν Οπότε πρόκειται για ένα ζήτημα επικοινωνίας και παρακολούθησης και συνέχειας που δόθηκε σε κάποια ζητήματα. Είναι βεβαίως το θέμα, το ερώτημα του πολίτη και το παρουσιάζει βεβαίως μια χαρά η έκθεση, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε το ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν και το τι είναι νόμιμο και τι όχι. Και βεβαίως αυτό είναι αυτονόητο πως έχει σημασία όταν αξιολογούμε τη συμπεριφορά της Κομισιόν απέναντι στον Μεσολαβητή. Γιατί η Κομισιόν η ίδια λυπάται για κάποια λάθη επικοινωνίας και οπωσδήποτε ο τρόπος αντιμετώπισης των ετοιμάτων του Μεσολαβητή δεν είναι ο βέλτιστος αλλά δεν παραβιάστηκε εδώ πέρα ο νόμος. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της διαδικασίας και του δικαιώματος του πολίτη για την ορθή λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πώς εκπλήρωσε η Κομισιόν της υποχρεώσεις της απέναντι στο κράτος μέλος. Σήμερα, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες, διαπιστώνουμε πως η Κομισιόν έκανε αυτό που ήταν εφικτό. Μάλιστα, αν δούμε πως υπήρχε λίγη κάποια ε, περιορισμένη αλληλογραφία, αλλά βλέπουμε πως οι περισσότερες ε, απαιτήσει ε, οι οποίες υπήρχαν εκπληρώθηκαν και αυτό σημαίνει πως αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος Μποστινάρου για άλλες περιπτώσεις της Επιτροπής ε, Αναφορών ότι δηλαδή το θέμα μας εδώ πέρα είναι όταν δεν πηγαίνει μια χαρά η ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναγκαστικά καταλήγουμε σε μια εξέταση ex post. Αυτό έγινε και μάλιστα συμπτωματικά γιατί υπήρχε ένα ακόμη μεγαλύτερο έργο που αφορούσε τον τρίτο διάδρομο έγινε μια ευρύτερη εξέταση στην περίπτωση αυτή δε όχι εξ αλλά ευθύς εξ αρχής και με τρόπο υποδειγματικό. Το τρίτο επίπεδο είναι τι έκανε το κράτος μέλος. Και εδώ πέρα δεν παραβιάστηκε πάλι το δίκαιο αλλά και εδώ πέρα ε, είναι ξεκάθαρη η έκθεση και σωστή επί της ουσίας γιατί πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα πως πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα διάφορα ζητήματα τα οποία παρουσιάζουν κάποιες ε, δυσαρμονίες γιατί οπωσδήποτε και ο Μεσολαβητής μας ζήτησε να μελετήσουμε αυτό το ζήτημα, να το αναλύσουμε. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πως η Κομισιόν σε αυτή τη φάση της έκθεσης έκανε τη δουλειά της με τρόπο πάρα πολύ θετικό και επικοδομητικό και η Επιτροπή μας σήμερα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο εδώ πέρα που ελπίζω να συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι ε, είναι σύνεπες και νομίζω μπορούμε να το υπερασπιστούμε ως Επιτροπή γιατί μας το επιτρέπει αυτό η ποιότητά του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έχετε το λόγο κυρία Ουκέν για το αν θέλετε να μας διευκρινίσετε για να θα έρθουν οι εκπρόσωποι των αρχών. Έχετε το λόγο κυρία Ουκέν. Ja, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κάποια λίγα σχόλια. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Νομίζω πως είχα μια επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή γιατί επιτύχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα με αυτό τον τρόπο. Έχω λίγα σχόλια. Γενικά, ε, σχόλια που αφορούν βεβαίως ε, την Κομισιόν και για το εάν η ερμηνεία είναι ευρύτερη ή στενότερη. Όσοι από ήμασταν βουλευτές σε εθνικά κοινοβούλια, εγώ ήμουν 20 χρόνια, συχνά ε, είχαμε κάποιες αιτιολογικές σκέψεις όπου λέγαμε ίσως να μην έχουμε λάβει υπόψη κάποια πράγματα και αντί να τα αναφέρουμε όλα, ε, θα ρίχνουμε τις αρχές να επιδεικνύουν κάποια φαντασία και κάποια κατανόηση επίσης. Και να μην ε, συμπεριφέρονται τυπολατρικά και να βασανίζουν τον κόσμο. Και νομίζω πως έχει δίκιο εδώ πέρα ο Μεσολαβητής. Ε, δηλαδή δεν ζητήσατε από την Αυστρία να επιδείξει μια τέτοια προσέγγιση. Γιατί οι πολίτες θα ήθελαν μία, όπως είπα, ανεξάρτητη αξιολόγηση. Γι' αυτό συμπεριέλαβα αυτή την κριτική ε, της Αυστρίας εδώ πέρα και την κριτική που άσκησε ο μεσολαβητής της Κομισιόν ε, όσον αφορά τον κύριο Μαρτίνες Μαρτίνες. Δεν είναι μεταφυσικό το ζήτημα. Η μεταφυσική για μένα πάει πολύ πιο πέρα από τη φαντασία, αλλά εντάξει, ίσως εδώ, και εδώ πέρα διαφέρουμε. Το άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες ε, αντιφάσεις και συγκρούσεις μεταξύ μας, αλλά εκπροσωπούμε και τους πολίτες όπως ακριβώς κάνει και ο Μεσολαβητής. Και θεωρώ πως η δικιά μας η δουλειά είναι να είμαστε λογικοί και γενναιόδοροι και να μην έχουμε πάντα τη στενή νομική ερμηνεία της νομοθεσίας. Ε, γιατί εδώ πέρα πρόκειται και για μια γκρίζα ζώνη, αν θέλετε. Αλλά νομίζω πως ο Μεσολαβητής έχει πιο δίκιο από την Κομισιόν. Αλλά βεβαίως γεγονός είναι πως τα πράγματα βελτιώνονται. για τον συνάδελφό μου, δε, τον κύριο Μαρτίνες. Δεν είχατε ακούσει τη συζήτηση την προηγούμενη φορά επί της εκθεσής Ματσόνη για τον Μεσολαβητή. Αλλά εκεί πέρα κατέστησε σαφές πως αυτό το οποίο αναμένουμε εμείς και ο Μεσολαβητής είναι πως το συντομότερο δυνατόν πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό, όχι κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμό για την ορθή διοίκηση και τη χρηστή διοίκηση και δεν μπορώ να πω πως ε, μας υποσχέθηκε κάτι τέτοιο ο Επίτροπος Σεύκοβιτς. Μάλλον τον ευνηδιάσαμε με το αίτημα αυτό και στην έκθεση Μασόνη και στα σχόλιά μας ε, στη συζήτηση. Αλλά ο Επίτροπος είπε πως ε, εντάξει, ίσως είχαμε κάποιο δίκαιο. Οπότε πηγαίνετε, απευθυνθείτε στον κύριο Επίτροπο και στους άλλους επιτρόπους, πείτε τους πώς χρειαζόμαστε τον κανονισμό αυτό το στομότερο δυνατόν. Για να ξέρουμε πώς ορίζεται η σωστή διοίκηση, η χρηστή διοίκηση, γιατί αυτά αναφέρονται και στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη χάρτα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποφεύγουμε τη διαφάνεια και με τρόπο τόσο δημιουργικό κιόλας. Αλλά σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Συμφωνώ πώς θα μας βοηθήσει το θέμα αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μπρέκλεντ, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Για το τελευταίο σημείο να σας πω ότι ε, σε σχέση με τον κανονισμό αυτό ασχολείται ε, και θα ο οργανισμός. Ε, θα μεταφέρω βέβαια το μήνυμά σας και στον Επίτροπο Σεύκοντιτς. Κατόπιν να δώσω το λόγο στην κυρία Ουσούλα Χαουπνέρ, ε, η οποία είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Αυστρικής Αντιπροσωπείας Αναφορών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά κυρίως κυρίες και κύριοι βουλευτές μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Σας ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση εξ ονόματος της αντιπροσωπείας μου για το ότι μπορούμε σήμερα να παρακολουθήσουμε την συζήτησή σας και να δούμε τα σημαντικά θέματα που αποτελούν την δραστηριότητα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή το να, ακούνε, να ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανησυχίες των πολιτών. Εμείς είμαστε μια αντιπροσωπεία που αποτελείται από τέσσερις ε, προέδρους ε, ομάδων ε, που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πράσινη ομάδα για λόγους ανηλυμένων υποχρεώσεων απουσιάζει, αλλιώς θα ήμασταν πέντε ομάδες εδώ πέρα και βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα για να λάβουμε αφενός πληροφορίες ε, και για να ανταλλάξουμε εμπειρίες για το πώς ε, ε, υπάρχει, αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Χαιρόμαστε επίσης για το ότι σήμερα στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο αναφορές από την Αυστρία. Το ένα ήταν το αεροδρόμιο της Βιέννης το οποίο συζητιέται ήδη και ένα άλλο ζήτημα το οποίο, με το οποίο ασχολείται η συνάλφος Άννα Χέλερα ε, πρόκειται για ένα γεωργικό ε, ζήτημα νομίζω θα το δείτε το απόγευμα το δικαίωμα του αναφέρεστε στις αρχές είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Αυστρία όπως ε, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι δικαίωμα που ασκούν πάρα πολλοί πολίτες. Στην Αυστρία έχουμε την ε, εμπειρία πως ε, ειδικά σε καιρούς όπου ο κόσμος είναι πιο επιφυλακτικός απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς ε, και πέρα που αμφιβάλλουν για την ικανότητα ε, των πολιτικών και της πολιτικής προσφεύγουν περισσότερο στο μέσο των αναφορών ε, και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πολιτών έχουν δηλαδή αυτό το μέσο της άμεσης δημοκρατίας και για προσωπικά τους ζητήματα αλλά και για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Γι' αυτό και στην Αυστρία θεωρούμε πως ε, η Επιτροπή Αναφορών είναι πάρα πολύ σημαντική για να ακούγεται η φωνή των πολιτών και πρέπει να τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ως ένα φόρουμ έκφρασης της πολιτικής βούλησης και πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί και βεβαίως είναι σημαντικό να παραμεριστούν διάφορα εμπόδια γραφειοκρατικής φύσης, οικονομικής φύσης, έτσι ώστε να είναι απλούστερη η πρόσβαση. Ελπίζουμε επίσης σήμερα στο πλαίσιο των συζητήσεών μας ε, να μάθουμε κάποια πράγματα για, την, για τις πρωτοβουλίες πολιτών που μας δίνουν νομίζω μια νέα ευκαιρία για να συνεργαστούμε και σε αυτό το επίπεδο και βεβαίως πρέπει να πούμε πως ε, και στην Αυστρία και σε άλλες πρωτεύουσες υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα για την γραφειοκρατία. Ε, ίσως και εδώ πέρα θέλουμε περισσότερη και ευκολότερη πρόσβαση γιατί θα πρέπει όπως είπα να μπορέσει να λειτουργήσει και στην πράξη αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών αλλιώς θα αποτύχει ευθύς εξ αρχής αυτή η πολύ καλή ιδέα δεν θα σπαταλήσω άλλο το χρόνο σας. Απλά να πω στο τέλος το εξής. Το δικαίωμα της, ε, του λόγου και της συναπόφασης ε, των πολιτών είναι μια σημαντική βάση για τη δημοκρατία. Έτσι ήταν πάντα και ελπίζω έτσι να συνεχίσει να είναι. Και Νομίζω πως η συμμετοχή αυτή των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει και στο μέλλον να παραμείνει νομίζω κεντρικό στοιχείο της ε, δημοκρατίας μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποδοχή σήμερα. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 12 Δεκεμβρίου και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2013. Τώρα περνάμε στην συζήτηση ε, των αναφορών που έχουμε στην ημερήσια διάταξη 7 αναφορά 759 του 2011 της Ελίζ Μισού με δύο υπογραφές που αφορά τις αντιδράσεις εναντίον ενός χώρου αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στο Ζουρονσό, ο οποίο κατά τα λεγόμενα παραβιάζει την οδηγία σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Η αναφέρουσα δεν είναι παρούσα, αλλά η Σαντρίν Μπελγή την αντικαθιστά, η βουλευτή Σαντρίν Μπελγή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. λόγω της απουσίας των αναφερουσών θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα διακυβεύματα αυτής της αναφοράς και μετά θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και να ακούσουμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να μας πει σχετικά με το φάκελο αυτό. από το 2009 χρονολογείται αυτός ο φάκελος, η εταιρεία Total στην κοινότητα Juronson πέτυχε μια άδεια για τον ενταφιασμό 100.000 τόνων διοξίδιο του άνθρακα ε, στο κέντρο ε, του Αμπελώνα που έχει ε, ονομασία προέλευσος και που σε μια περιοχή που είναι σεισμολογική είναι κατοικημένη η περιοχή. Τα τρία προηγούμενα έργα προγράμματα ήταν ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε στις κάτω χώρες και διακόπηκαν λόγω της αντίδρασης των τοπικών κοινοτήτων. Οι κίνδυνοι στους οποίου εκτίθεται ο πληθυσμός και η οικονομία του τόπου με διαρροή ε, και οξύδωση του υδροφόρου ορίζοντας, σεισμολογικός κίνδυνος που αυξάνεται ε, και υπάρχει κίνδυνος εισπνοής των προϊόντων αυτών από τους κατοίκους σα Σήμερα, τρία χρόνια μετά από το 2001, είμαστε στο 2012, μετά από αυτήν την άδεια που δόθηκα, μάθαμε ότι η εταιρεία Total σκέπτεται να κλείσει την εγκατάσταση αυτή και η βασική ανησυχία των αναφερουσών είναι το μέλλον αυτού του χώρου και τα διάφορα μέτρα που θα ληφθούν για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση ε, και η αποκατάσταση του χώρου αυτού, αλλά κυρίως η παρακολούθηση αυτής της αποθήκευσης και τα μέτρα ασφαλείας και των μέτρων Για Οι αναφέρουσε επίσης επισύρουν την προσοχή μας πάνω στο γεγονός ότι μέχρι τώρα η εταιρεία Total που διαχειρίζεται αυτή την αποθήκευση διοκισκηδίου του άνθρακο, ε, διατηνόταν ότι δεν έπρεπε να εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο και κυρίως την οδηγία 2009-31 για την αποθήκευση του του άνθρακος με βάση την αρχή ότι ήταν κάτω από την δυναμικότητα που προβλέπεται από το άρθρο 2.2 της οδηγίας αυτής που προβλέπει ότι η οδηγία ε, δεν ισχύει ε, ε, όταν πρόκειται για δυναμικότητα κάτω των 100 κιλοτόνων ενώ η απόφαση αναφερόταν σε 120.000 τόνους στην άδεια που μετά τροποποιήθηκε, δηλαδή μια δυναμικότητα αποθήκευσης ανώτερη που από ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 2.2 της Οδηγίας 2009-31 ε, και η εξαίρεση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Ε, πρόκειτο για ένα από τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντέτεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, εξαιρέσει ε, την εταιρεία Total από τα μέτρα παρακολούθησης για τα λόγους ασφαλείας λέγοντας ότι τα μέτρα, τα μακροπρόθεσμα είναι ευθύνη της εταιρείας και αυτή πρέπει να αποδείξει ότι τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στην εξαίρεση ενώ οι αναφέρουσες τώρα ε, ζητούν στην εταιρεία, εφόσον θα διακόψει την αποθήκευση, ζητούν από την εταιρεία και την Γαλλία να εξασφαλίσει η εταιρεία Total. Δεν θα φύγει έτσι απλώς, αλλά ότι θα λάβει όλα τα μέτρα παρακολούθησης του χώρου αυτού μετά ε, το κλείσιμο της εγκατάστασης αποθήκευσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δώνω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Γεφσεβιαντικό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε στη συνεδρίαση αυτή. Όπως ε, δηλώσατε και εσείς, η Κομισιόν ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η αίτηση, αυτή η αναφορά αφορά μια παράμετρο για αποθήκευση 90.000 τόνων και δηλαδή είναι κάτω από τα όρια των 100.000 τόνων αυτό το όριο των 100.000 τόνων αποτελεί το πεδίο της ε, οδηγίας 2009-31 το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής και για αυτό το λόγο δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί στο ζήτημα αυτό γιατί σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας αυτό είναι ένα θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα κατόπιν επικοινωνίας με τις γαλλικές αρχές ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2009-31 της Κυρία Μπελιέ, Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Θέλω απλώς να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών να κρατήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθυνθεί στο γαλλικό κράτος και στην εταιρεία Total και να ζητήσει να μας παρουσιάσουν την κατάλληλη τεκμηρίωση, να μας διασφαλίσουν ε, ότι ε, θα υπάρξει παρακολούθηση για το τι γίνεται σε αυτή την τοποθεσία. Όπως σας είπα, πρόκειται για αποθήκευση δεξιδίου του άνθρακα. Θα υπάρχουν και μικροπρόθεσμες συνέπειες. Ε, ακούσαμε ότι κάτω από τις 100.000 τόνους δεν είναι αρμόδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως υπενθυμίζω ότι η αρχική άδεια ήταν για 120.000 τόνους και υπάρχει διάταγμα τροποποίησης και μειώνει το ποσό αυτό στους 90.000 τόνους. Δεν ξέρουμε ακριβώς όμως ποιο είναι το ποσό αποθήκευσης ε, που αποθηκεύτηκε τελικά και αν ε, δεν έχει αρμοδιότητα η Κομισιόν για την εποπτεία αυτής της τοποθεσία, νομίζω ότι η δική μας ε, ευθύνη ως Ευρωβουλευτές είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέτρα θα ληφθούν από την εταιρεία κατόπιν σύσταση του γαλλικού κράτου για να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων. Ο κύριο Μαρτίνε Μαρτίνε. Ναι, πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι τα όσα λέει η κυρία Μπελιέ είναι απόλυτα λογικά. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να συνεχίσει η ανοιχτή αναφορά, μέχρι τουλάχιστον να έχουμε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες ε, που θα μας ταλούν από τις γαλλικές αρχές. Δεν ξέρω αν η ίδια η εταιρεία απευθεία δίνει πληροφορίες ή όχι, αν θα τις δώσει μέσω των αρμοδίων αρχών, ε, που είναι ο δικός μας συνομιλητής. Όμως εμένα, όπως και να έχει, μου φαίνεται λογικό και αρκετά ανησυχητικό το θέμα, έτσι ώστε να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Παρακαλώ, κύριος Γιάννη. Ο κύριος Γιάννη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Μα κοιτάξτε, οι, οι τιμέ τιμές είναι, είναι αυτές που είναι. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτή είναι η οριακή τιμή. Ζητώ όμω να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά για να δούμε ακριβώς πόσο είναι το, το ποσό που αποθηκεύεται. Γιατί εδώ πέρα έχουν δίκιο οι αναφερόμενοι. Δεύτερον, ακόμα και αν δεν είμαστε αρμόδιοι, το εξετάζουμε ακόμα, αλλά ακόμα και αν δεν είμαστε αρμόδιοι, πρέπει οπωσδήποτε και η Γαλλία να, να τηρεί την περιβαλλοντική ε, νομοθεσία. Δηλαδή όχι όταν ασχολείται η Ευρώπη κοιτάνε το τι γίνεται με το περιβάλλον και άμα δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμιά σημασία, δεν είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό θα πρότεινα να ενημερώσουμε τους ε, πολίτες εδώ πέρα να δουν και στο Παρίσι τι γίνεται γιατί είναι και εθνική υπόθεση δηλαδή και να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά να δούμε όντως πόσο θα ε, αποθηκευτεί εδώ πέρα και να απευθυνθούν νομίζω και στη Γαλλική Επιτροπή Αναφορών Γιατί είναι, είναι και, και εθνική η αρμοδιότητα, δεν τίθεται ζήτημα. Ταιριάζει με αυτό το οποίο είπα και πριν ε, για την Αυστρία, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε η Επιτροπή Αναφορών με τα κράτη-μέλη όταν δεν ξέρουμε ποιος έχει ακριβώς την αρμοδιότητα, ακριβώς για αυτό το οποίο είπα. Τις εθνικές ή περιφερειακές επιτροπές αναφορών. Νομίζω πως εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα, ένα μέρο του προβλήματο, δηλαδή, ε, πρέπει να το επιφορτιστεί και η Γαλλική Ανάλογη Επιτροπή. Ο κύριος Μποστινάρο έχει τον λόγο. Συμμερίζομαι πλήρως την ιδέα ότι πρώτα απ' όλα η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Δεύτερον, νομίζω ότι μπορούμε να προετοιμάσουμε μια επιστολή για την Γαλλική Εθνοσυνέλευση για να συζητήσουμε μαζί της ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δύο επιτροπές, η δική μας η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν ξέρω αν ακριβώς υπάρχει μια αντίστοιχη επιτροπή στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κάποιο όργανο το οποίο να είναι επιφορτισμένο με τέτοια προβλήματα, με τέτοια ευαισθησίας και πιθανόν ε, να έχουμε ένα διάλογο με την κυβέρνηση και τις γαλλικές αρχές για το θέμα αυτό που είναι ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο, αρκετά λεπτό, ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνει πειράματα και τεχνολογίες που βρίσκονται στην αρχή της βιομηχανικής του σταδιοδρομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάρ, θα ήθελα επίσης να σας δώσω μια πληροφορία. Δεν υπάρχει Επιτροπή Αναφορών στην, στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, προτείνω να είναι η δική μας Επιτροπή που να ζητήσει από τις γαλλικές αρχές διευκρινήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε εμείς στις αναφέρουσες. Υπό το φως των όσων παρουσιάστηκαν θεωρώ Δεδομένου των όσων παρουσιάστηκαν, νομίζω ότι αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ούτω ώστε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυ. Τώρα περνάω ε, στο σημείο 8, αναφορά 385-2011 της Νόουλιν Μακμάνου, εξ ονόματο της οργάνωσης SWAP, σχετικά με οικοδομικό έργο σε περιοχή που εικάζεται ότι εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στην Κομιτεία ε, Wicklow είναι παρούσα η αναφέρουσα και θα μας κάνει μια παρουσίαση με PowerPoint. Good morning, ladies. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι, γιατί κάποιες ε, διαφάνειε ε, που έστειλα πριν δεν έφτασαν, είχαμε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή. Θα ήθελα να παρουσιάσω την κοινότητα που εκπροσωπώ πρόκειται για ε, μια παράκτη πόλη στην ανατολική ακτή της ε, Ιρλανδίας ε, και ο ποταμός Ντάγκολ περνά από το κέντρο της πόλης μου και βρίσκεται και είναι κατοικημένη η βόρεια περιοχή του ποταμού. Η δική μας γειτονιά είναι μια μικρή λεκάνη γης και έτσι λοιπόν όταν έχουμε πάρα πολλές βροχές και χαμηλή πίεση υπάρχουν ε, πλημμύρες ε, και καθώς έχουμε πολύ υψηλό ε, ποσοστό ηλικιωμένων και ανθρώπων με που ζουν στην περιοχή μας γενικά έχουμε ισόγεια σπίτια και αυτό αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Η Βίλα Μαρία Παρκμητός είναι ένα από τα δύο κέντρα για ανθρώπους με ψυχικές νόσους και βρίσκεται 250 μέτρα από το ποτάμι. Είχαμε πολλέ καταστροφικές πλημμύρες το 1995 ε, το, το 1931, το 1966, δηλαδή κάθε 20 με 30 χρόνια βλέπουμε πλημμύρες και το 2005 η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ ημών και της θάλασσας ε, εκεί ε, πυκνοκατήθηκε και η τα νερά της πλημμυράς που έρχονται από το νότο όταν υπερχειλίζει το ποτάμι και από τα δυτικά περνούν από τα δικά μας σπίτια όταν πηγαίνει άναντι το ποτάμι και υπερχειλίζει. Έτσι βλέπετε εδώ πως μοιάζει η γη ε, και τι έγινε όταν είχαμε τις πλημμύρες τον Αύγουστο του 1966. Βλέπετε εδώ κάποιους εθελοντές πολιτικής άμυνας ε, ε, προσπαθούσαν ε, εκεί να σώσουν κάποιους ανθρώπους προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους και το ίδιο και εμείς και έφτασαν τις, ε, οι πλημμύρες μέχρι και δύο μέτρα τα νερά γύρω στις 4 η ώρα αλλά σταμάτησαν ε, μέσα σε ώρες ε, να έρχονται τα νερά γιατί ουσιαστικά συνέχισαν την πορεία τους όπως πάντα. Ο δρόμος που βλέπετε άνοιξε στα δύο από τη δύναμη του νερού από τη δύναμη της πλημμύρες και άρχισε κάποιοι ζήτησαν άδεια 2,2 ε, εκατομμυρίων για οικιστικά σχέδια. Εμείς ε, Βλέπουμε εδώ τι προτείνουν να κτίσουν στην περιοχή που μόλις είδατε. Είχαμε κάποια ε, σοκινηματογράφους, ε, εστιατόρια ε, που θα τα έκτιναν σε εφταόρφο κτίριο. Έτσι λοιπόν δημιουργήταν ε, ένα φράγμα γύρω από την πεδιάδα ε, γιατί ουσιαστικά θα έφτανε το κτίριό του στα 7 μέτρα. Η δικαιολογία που δόθηκε από τους πολιτικούς μας ε, και ε, αυτό ήταν κατά την ανάπτυξη της Ιρλανδίας είναι ότι ε, θα υπήρχαν αντιπλημμυρικές υποδομές για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο. Εμείς ποτέ δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης στα 47 ε, εκτάρια της περιοχής. Απλώς ζητάμε να επιστραφούν σε έναν ασφαλή χώρο ε, και τα 19 εκτάρια πίσω από αυτά να αναπτυχθούν οικιστικά. Αντίστοιχα είχαμε κάποια επιτυχία. Η πρώτη αίτηση απορρίφθηκε όταν κάναμε ένσταση στον αρμόδιο φορέα σχεδιασμού και τώρα διπλημμυρικές υποδομές ε, στείνονται από την πλευρά του ποταμού και πληρώνονται ε, από δημόσια ε, κονδύλια και όχι από ιδιωτικούς επενδυτές όμως. Ε, υπήρξε και μια δεύτερη αίτηση και πάλι αποφάσισε το Συμβούλιο να απορρίψει τη Συμβουλή των Επιθεωρητών και έδωσε μια άδεια δεκαετή για οικοδόμηση σε αυτή τη ζώνη από τον Ιούνιο του 2010. Μέχρι τότε ε, υπήρξαν οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επενδυτές ε, και ήδη ε, όταν έσκασε η φούσκα οικιστική στην Ιρλανδία ανέλαβε το δημόσιο. Έτσι λοιπόν τώρα αυτή η γενική στους πολίτες και όχι στους συνδιώτες όμως αν δεν αλλάξει η οριοθέτηση της περιοχής, τότε θα έχουμε και ανθρωπιστική και οικονομική καταστροφή. Και σε μεγαλύτερο κίνδυνο θα είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι και άνθρωποι με αναπηρίες. Το είδαμε αυτό στην Εορλεάνη το 2005, όταν ήρθαν ε, οι περιορισμοί για την οικοδόμηση και ε, είχαν παραμεληθεί δραστηριότητες συντηρήσεις ε, των κτηρίων. Δεν υπάρχουν ε, οι πόροι από εμά για να προσφύγουμε στα δικαστήρια στην Ιρλανδία. Έτσι λοιπόν ήρθαμε στην Ευρώπη για να ε, ζητήσουμε δυνάμει τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το δικαίωμα τη ασφάλεια ε, των ανθρώπων, το δικαίωμα σεβασμού απέναντι στα σπίτια μα, το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου και το δικαίωμα των ηλικιωμένων και των ανάπηρων γειτόνων μα να είναι προστατευμένοι, το δικαίωμα στην αηφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία και πάνω απ' όλα το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια και όσων ε, απειλούνται από την ε, χωροταξία σε αυτή την περιοχή. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν ε, χρειαστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταστήσουν πραγματικότητα τα ιδανικά που αναπτύσσονται σε αυτή τη χάρτα και να βρούμε επιτέλους τη δικαιοσύνη που επιζητάμε από το 2005. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε για αυτήν την ε, λεπτομερή παρουσίαση και τώρα δίνω τον λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Επιτροπής, τον κύριο Μπρέικλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συζήτηση για την αρχή της επικουρικότητας και ένα από τα σημεία κλειδιά σε αυτή την περίπτωση είναι η οριοθέτηση, η χωροταξία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, η απόφαση αυτή για την οριοθέτηση των ζωνών ε, χωροταξικά δεν εμπίπτει το θέμα αυτό ε, στον νόμο των ευρωπαϊκό στην νομοθεσία την ευρωπαϊκή. εξατάζουμε ε, την ε, οδηγία για τις πλημμύρες ε, που εγκρίθηκε μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Ευρώπη, αλλά εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία υποβάλλονται σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που πρέπει να κατατεθούν μέχρι τα τέλη του 2015. Ε, μια αναφορά ε, ε, απορρίφθηκε της κυρίας Νόλεν Μακνάνο, στη δεύτερη φορά έγινε παραδεκτή και εξετάσαμε τα θέματα των πλημμυρών. Νομίζω ότι αναφέρουσα δεν, δεν συμφωνεί με την περίπτωση αυτή. Θα πρέπει η Κομισιόν να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η κανονική οδός θα ήταν η προσφυγή στο δικαστήριο διότι η λύση θα ήταν να αμφισβητήσει κανείς την απόφαση πενόλα στα δικαστήρια. Υπάρχουν μερικά προβλήματα ως προς το χρόνο, τις προθεσμίες. Ξέρουμε ότι η πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ανοιχτή περίπτωση σχετικά με την Ιρλανδία για την πρόσβαση στο δικαστήριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θα έλεγα ότι σε σχέση με την οδηγία περί των πλημμυρών δεν υπάρχει λύση ε, σχετικά με την ε, οδηγία για την αξιολόγηση αντικτύπου στο περιβάλλον επίσης και η προσφυγή στο, στο, στα δικαστήρια της Ιρλανδίας με διαδικασία επί είναι μια οδός. Σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες ε, βλέπω ότι γίνονται έργα ε, για την συγκράτηση των ε, πλημμυρών, των υδάτων. Έχουμε επίσης μια διαδικασία επί παραβάση κατά της Ιρλανδίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα έργα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. Αναφέρατε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δυστυχώς ε, συζητείται πάρα πολύ συχνά ο χάρτης αυτός εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Οι υποχρεώσεις του χάρτη για τα κράτη-μέλη είναι μόνον όταν εφαρμόζουν ε, νομοθεσία ευρωπαϊκή. Αυτά είναι τα όρια, οι περιορισμοί του άρθρου 51. Οι διατάξεις λοιπόν του χάρτη αυτή ε, εμπλέκουν τις, τα ευρωπαϊκά όργανα μόνο όταν πρόκειται για ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, γι' αυτό ασχολείται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης εδώ. Ε, δεν εφαρμόζεται ευρωπαϊκός νόμος, αλλά ε, Ιρλανδικός νόμος. Μόνο όταν εφαρμόζεται ευρωπαϊκός νόμος υπάρχουν οι υποχρέωσεις του χάρτη. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω ένα μέσο από ευρωπαϊκής απόψεως για να ασχοληθούμε με τις δυσκολίες σας. Νομίζω ότι για την ώρα το πρόγραμμα αυτό, το οικοδομικό έργο αυτό δεν έχει κτιστεί. Ε, ε, ε, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πρόσβαση στις πληροφορίες για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα όρια και περιορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνω τον λόγο στον Πάουλι Μέρφυ, συναδελφό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Καολίν για την παρουσίασή της. Αυτό το οποίο έχουμε σε αυτή την περίπτωση και το είδαμε την Ολύν είναι μια μικρογραφία των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ιρλανδία τα τελευταία 10-15 χρόνια όπου τα συμφέροντα των εργολάβων ήταν αυτά τα οποία προηγήθηκαν όλων των άλλων. Και εδώ πέρα έχουμε έναν εργολάβο ο οποίος ε, υπερήξει όχι μόνο του δικαιώματος στην ποιότητα ζωής των απλών ανθρώπων αλλά και πιθανώς ε, του δικαιώματος της ζωής μιας ε, κοινότητας ε, κυρίως ηλικιωμένων και εργαζομένων. Και αυτό το οποίο γίνεται με αυτή την καμπάνια είναι πως οι απλοί άνθρωποι υψώνουν το ανάστημά τους στους εργολάβους και τους πολεμάνε σε κάθε τους βήμα κτλ. Αυτό έχουμε. Και είναι απίστευτο. Υπό την έννοια πως δεν είναι πως η πολεοδομία δεν είχε χάρτες ε, για τον κίνδυνο πλημμύρας. Υπήρχε κίνδυνος πλημμύρας, αλλά μετά την ε, σχεδίασαν ε, για περιοχή κατοικίας υψηλής πυκνότητας. Και βαρκεί να δείτε το βίντεο για να δείτε το τι μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι μία από τις τέσσερις πλημμύρες τον αιώνα που μας πέρασε και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση μπορεί να οδεύουμε σε μια τέτοια πάλι παρόμοια πλημμύρα και βεβαίως αν χτίζονταν αυτά τα κτίρια και η λεκάνη αυτή πλέον απορροήσει, θα υπήρχε και θα είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό το οποίο λέει η Νολίν για την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι σωστό το δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ηλικιωμένων, μη διακριτική μεταχείρισης, δικαίωμα στη ζωή κτλ. Αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε αυτή την κοινότητα να αντισταθεί στους εργολάβους. Αυτό το οποίο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και αν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψη στην Ιρλανδία ναι, αν μπορούσαμε να επισκεφτούμε και τον Μπρέι θα ήταν, ε, θα ήταν εξαιρετικό γιατί όπως και με το βίντεο μόνο εάν το δούμε θα αντιληφθούμε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό το, το, το έργο. Γιατί μπορεί να νικήσει εδώ πέρα η κοινότητα ακριβώς γιατί πλέον ε, ε, είναι δημόσια αυτή η έκταση Οπότε είναι πλέον στα χέρια των, των φορολογουμένων. Οπότε τουλάχιστον δεν θα πρέπει να γίνει ε, η ανοικοδόμηση και όταν μετά ξαναγίνει πολεοδομικός σχεδιασμός σε κάτι χρόνια να, να ξαναδούν το, το ζήτημα της περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρότεινα να αφήσουμε, κύριε Μέρφη, ανοιχτή την αναφορά, να ξαναδούμε το ζήτημα με τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή Αναφορών της Ιρλανδίας, ίσως του χρόνου να προγραμματίσουμε και μια επίσκεψη για να το δούμε και με τι οπικέ αρχές. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σωστά είπατε Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών στην Ιρλανδία, αλλά έχετε δίκιο. Ε, μπορούμε λοιπόν να τους ζητήσουμε και πληροφορίες. Ε, εντάξει, η ανθρώπινη λογική θα έλεγε πως δεν χτίζουμε σε μια τέτοια περιοχή, αλλά καμιά φορά βεβαίως συμβαίνει. Εμένα με, με ενοχλεί ε, αφενός βλέπω πως μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχει μεταφερθεί και εφαρμοστεί η οδηγία και άρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος πλημμύρας. Μα θα έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μπορούμε να τους ρωτήσουμε. Έχουμε μία αναφορά. Ισχύουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι άνθρωποι ή εσείς ξέρετε κάτι διαφορετικό και θα μας πούνε. Γιατί δεν, δεν είναι ικανοποιητική εδώ πέρα η κατάσταση. Γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα θέλουν να αποτρέψουν και, και ζημία των ε, φορολογουμένων. Εάν οικοδομηθεί αυτή η περιοχή, ε, δεν είναι και, λογικό αυτό το πράγμα, πράγματι να συμβεί. Οπότε ζητάω να απευθύνουμε μια επιστολή στην Επιτροπή Αναφορών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και μια, μια απάντηση για το ποια είναι, η αλήθεια, έτσι, τι συμβαίνει όντως. και να δούμε μετά τι θα γίνει. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, να μην ανοιχτή αναφορά. Δεύτερον, ναι, να στέλνει μια επιστολή στις αρχές της Ιρλανδίας για να μας δώσουν και τη δική τους αξιολόγηση. Γιατί ε, ουσιαστικά το προπετούμενο είναι η άδεια οικοδόμησης και αν εκδόθηκε με τέτοια άδεια με ποια νομική και τεχνική βάση εκδόθηκε. Και εδώ βλέπουμε ότι εμπλέκονται και πολλά άλλα σχέδια από ε, την κοινότητα μέχρι τους μελλοντικού ιδιοκτήτες αυτών των ε, εγκαταστάσεων αυτών των κτηρίων είναι σημαντικό να λάβουν οι άνθρωποι αυτοί απαντήσει από τι ελληνικέ Αρχέ. Και θα πρέπει αυτό το θέμα να είναι στην ημερήσια διάταξή μα όταν ε, η δική μα ε, αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί την Ιρλανδία. Σα ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Μπουστινάρου. Αυτό θα πράξουμε. Θα στείλουμε μία επιστολή στι Ιρλανδικέ αρχέ, ε, προκειμένου να ζητήσουμε περαιτέρω εξηγήσει, κυρία Όκεν. Πολύ σύντομα Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν και μια μικρή παρατήρηση ε, στη συνεχιζόμενη ε, μάχη που δίνουμε με την Κομισιόν ε, για το θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ή να αποκλείσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί ξέρουμε αυτή την παράγραφο από αυτήν την παράγραφο της χάρτας δεν είναι το δικό μας καθήκον να το διερευνήσουμε αν ένα ζήτημα αν δεν παραβιάζει την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποτελούν την απόλυτη βάση της συνθήκης. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο η Κομισιόν απλώς ε, να μας λέει πρέπει να πάτε πίσω στην επίπεδο για μένα είναι εξοργιστικό ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε κι εμείς ότι οι πολίτες της Ιρλανδίας δεν εκτίθεται σε έναν ε, τόσο ανόητο τρόπο χρήσης της γης. Και θα αναφερθώ και στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί για την οικονομία και το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα μιας ε, οικονομίας κοντόφελμπης ακόμη και μεσοπρόθεσμα θα αποδειχτεί πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι ένας οικονομικός τρόπος να σκεφτόμαστε αυτός. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν ξέρουν ε, καθόλου τι γίνεται στον κόσμο. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα, αλλά σας παρακαλώ πρέπει και λένε ότι εντάξει μπορούμε να το κάνουμε έτσι, μετά δεν θα υπάρχει κανένα αντίκτυπο, αλλά δεν είναι πιθανό αυτό. Η αναφέρουσα θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, ναι. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και που μας ακούσατε. Εμείς ε, ε δώσαμε αυτόν τον αγώνα κατά μιας πολύ μεγάλης εταιρεία με πάρα πολλά χρήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα και ένας ε, από τους λόγους που πιστεύω ότι αυτό το τρελό σχέδιο πέρασε ήταν ε, επειδή πραγματικά είχαν θράσος, ε, ήταν ε, τόσο τρελό, επομένως συνέχισαν να πιστεύουν κάποιοι ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος λόγος όμως. Ένα τετράχρονο παιδί δεν θα έκανε το ίδιο αυτό λάθος των πολιτικών που έδωσαν την άδεια, όμω προφανώ οι πολιτικοί δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο Δεν καταλαβαίνω γιατί η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται μόνο σε εμά το δικαίωμα στη ζωή, στο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, όταν έχει ε, παραβιαστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως σίγουρα η χάρτα είναι ευρωπαϊκός νόμος, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια, στο σεβασμό του σπιτιού του. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο στη δική μας κοινότητα. Και θα ήθελα επίσης να εξηγήσω ότι ε, με τις αντιπλημμυρικές υποδομές, ε, αν ο όγκος του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλος και σπάσουν οι αντιπλημμυρικές υποδομές, ή αν ε, δεν συντηρηθούν αυτές οι υποδομές ε, και ξέρετε ε, ο δικός μας Δήμος συχνά δεν συντηρεί, τότε υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος γιατί αν σπάσουν ανάντι οι υποδομές δεν μπορούν να ξανά χτιστούν και αν κάτι ε, οικοδομηθεί κατά του ποταμού ότε μιλάμε ε, για ένα πάρα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή περιοχή, 8 εκτάρια. Αν κάτι λοιπόν χτιστεί κατά αντί του ποταμού θα γίνουμε λίμνη και όλο αυτό το νερό θα έρθει στα σπίτια μας και θα μείνει στα σπίτια μας και δεν θα υπάρξει καμία αποζημίωση που να μπορεί να αντικαταστήσει τις ζωές που θα χαθούν ε, ε, δύο φορές έχει πλημμυρίσει το δικό μου σπίτι και είδα τα νερά να έρχονται μέχρι την πόρτα μου και αποζημιώθηκα γιατί έχω ασφάλεια άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν ε, να ε, ασφαλιστούν γιατί βρισκόμαστε σε μια τέτοια πλημμυρική περιοχή. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να τα σκεφτείτε όλα αυτά και σας ευχαριστώ. Νο, σας ευχαριστούμε και εμείς κυρία Μακμάνος. Συνεχίζουμε με το σημείο 9 αναφορά 1311-2010 του Αλεχάνδρου Σάντσες Γκαρσίας εξ ονόματος του Δήμου Λίνεα la Κονσεψιόν σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οικιστικού έργου στο Γιβραλτάρ. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον κύριο Ντρέκλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε υποβάλει ενδελεχείς εξηγήσει γιατί ε, δεν υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση παράβαση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, Βεβαίως το Σεπτέμβριο πέρσι έγινε έρευνα, ελέγξαμε ε, την ποιότητα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ελέγξαμε τις επιπτώσεις πάνω στα ισπανικά ύδατα κατά τη διάρκεια της ε, οικοδομής, της οικοδόμησης. Ορισμένα μέτρα υιοθετήθηκαν ούτως ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή. Ε, βεβαίως το έδαφος που χρησιμοποιούν το υπήρχε από τη δεκαετία του 1990 είχαμε ε, δύο ε, δυσμενείς επιπτώσεις ε, σε χώρους σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε και με τις αρχές του Γιμπραλτάρ δεν υπάρχουν επιπτώσεις σε χώρο που βρίσκεται αρκετά μακριά από την, το οικιστικό πρόγραμμα. Ξέρω ότι υπάρχει μια διαμάχη σχετικά ε, ανάμεσα για τον ε, ορισμό σχετικά, τον ονομασία ανάμεσα στο Γιβραλτάρ, ε, στις για το Γιβραλτάρ ανάμεσα στις Ισπανικές Αρχές και το Ηνωμένο Βασίλειο, όποιος όρισε την περιοχή. Αυτό όμως δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουμε ορισμένου ισχυρισμούς στην Λαλίνε Αντελακονσεψιόν ότι χάνεται άμμος από τις παραλίες και λάβαμε ε, από τις αρχές των Ηνωμένου Βασιλείου απάντηση σχετικά με την απώλεια άμμου. Δεν υπάρχει απώλεια και όλα τα στοιχεία, ε, λάβαμε όλα τα στοιχεία και ζητήσαμε από τις αρχές του Γιβραλτάρ που απήντησαν εδελεχώς και δεν, ε, δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κάποια παραβίαση του ευρωπαϊκού νόμου. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Ε, παρουσιάστηκαν διάφορα στοιχεία από την Κομισιό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε το θέμα αυτής της αναφοράς, αν συμφωνείτε. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη για την, στην Ιταλία από τις 29 στις 31 Οκτωβρίου θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών που συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη. Αρχίζουμε με την κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Μα εγώ την χάρη να μόνη παρούσα η οποία ήταν ε, τακτικό μέλος της αντιπροσωπείας. Της αντιπροσωπείας ήμασταν δύο, η άλλη ήταν η Judith Mavis, η οποία τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Οπότε θα κάνω κάποια πρώτα σχόλια. Σκοπός της επίσκεψης ε, ήταν ε, συνεχείς μας ανησυχίες για την ε, συνεχιζόμενη κακοδιαχείριση ε, της διαχείρισης αποβλήτων στην ε, Ισπανία. Εδώ και χρόνια αγνοούνται αυτά τα πράγματα και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν είναι καλή στην Ιταλία έχει καμιά φορά την πως όλη αυτή η σχετική νομοθεσία είναι επιστημονική φαντασία για τις Ιταλικές αρχές. Πριν λοιπόν να πάμε ε, αποφάσισε η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία παραβάση στο ΔΕΚ ε, κατά της Ιταλίας για να πληρώσει πρόστιμο η Ιταλία για τη μη συμμόρφωσή της και έχει κανείς την εντύπωση πως προτιμάει ο κόσμος εκεί πέρα να πληρώνει πρόστιμα από το να κάνει κάτι. Τι να πω, προτιμάει τις κυρώσεις. Είχαμε όμως μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη. Ήταν πολύ έντονο το ταξίδι μας. απασχόλησε και την κοινωνία και νομίζω πως είχαμε και κάποια θετικά αποτελέσματα. Δεν ήταν μόνο ζήτημα του σκανδάλου, αλλά ίσως βελτιωθεί κάτι στο μέλλον. Είχαμε μια συνάντηση την οποία παρακολούθησε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κλινή, ο οποίος γνώριζε το ζήτημα και το που πρέπει να καταβληθεί κάποια προσπάθεια και είπε πως δεν πρέπει να ε, ανεχτούμε κάτι τέτοιο αλλά βεβαίω είχαμε και εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ήταν σαφές πως ένα από τα βασικά ζητήματα στην Ιταλία είναι η διοίκηση και ζητώ συγγνώμη από τους Ιταλούς ε, συναδέλφους, αλλά είναι χάος. Πρέπει να μπορούμε να λέμε ποιος είναι ο υπεύθυνο και να έχει κάποιος την ευθύνη. Και προσπαθούσε ο ένας να το ρίξει στον άλλον. Όχι δε φταίω εγώ, είναι ο άλλος και από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή, η κατάσταση ήταν αστεία αστεία γελούσαμε για να μην κλάψουμε. Την επόμενη μέρα είχαμε δε μια συνάντηση στην Άπολη Ε, κόντεψα να πέσω από την καρέκλα μου. Γιατί ο Υπουργό Περιβάλλοντος της Περιφέρειας είπε πως είχαν 551 δημάρχους στην Καμπανία. 551 δήμαρχοι στην περιφέρεια. Οπότε βεβαίως δεν θα συμβεί τίποτα αν δεν έχουν οι πολίτες δυνατότητα να βρουν τον υπεύθυνο και πώς ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Πρέπει να το πούμε αυτό στην έκθεση είχα ότι και αυτή η κατάσταση ε, δηλαδή πρέπει να το γράψουμε και στην οδηγία χρειάζονται καλύτερη διοίκηση στην Ιταλία. Για να μπορεί να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα. Η επίσκεψή μας τώρα που πήγαμε, πήγαμε στη Μαλακότα, είδαμε τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν ε, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση όπως την πρώτη επίσκεψη που είχαμε άμεση επαφή αλλά αυτό το οποίο είδαμε στη Μαλακώτα μια τεράστια περιοχή ε, διαχείρισης αποβλήτων ε, ήταν απόβλητα στα οποία δεν είχε γίνει ακόμα διαλογή φτάνουν εκεί πέρα σε ένα εργοστάσιο σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και ως άνθρωπος βεβαίως δεν μπορεί κανείς να δει τι είναι μέσα στη μαύρη της σακούλα των σκουπιδιών εμείς στη Δανία δεν έχουμε μαύρες σακούλες, είναι διάφανες σακούλες. Και ποια ήταν η πρώτη επεξεργασία, τα βάζανε σε ένα μηχάνημα θρηματισμού και μετά κανα διαλογή. Μα χωρίς διαλογή και χωρίς να ξέρουμε τι είναι μέσα στις σακούλες τι κάνανε. Επίσης ήταν σαφές και στο Λάτσιο και στην Καμπανία πως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα υγείας τα οποία δεν τα έχουν πάρει σοβαρά εκεί πέρα. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη σαφήνεια για, το, για τα προβλήματα υγείας. Ένα από τα μέρη επίση που επισκεφθήκαμε ήταν το ΆΜΑΚ, όπου υπήρχε φόβερη δυσοσμία ή δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και το άσθημα μου. Ε, εν πάση περιπτώσει η, η δυσοσμία δεν βλάπτει την υγεία, αλλά βλάπτει την ποιότητα ζωής, όπως και ο θόρυβος. Αν υπάρχει συνεχής δυσοσμία, ε, βλάπτεται η ποιότητα ζωής. Όπως ε, και το να ζει κανείς σε μια περιοχή με θόρυβο. Και πρέπει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η δυσοσμία. Οι ε, αιτούμενοι θεωρούν πως προέρχεται από τη μεγάλη εκεί περιοχή κομποστοποίησης. Οι αρχές λένε πως η δυσοσμία προέρχεται από ένα εργοστάσιο αποτέφρωσης. Ε, πρέπει να βρουν από πού έρχεται όμως. Τέλος, να πω πως την τελευταία μέρα, δηλαδή την Τετάρτη που μας πέρασε στην Άπολη, είχαμε μια συνάντηση η οποία ήταν επιτυχής. Ήταν παρόντες ε, πολλοί από τους αναφερόμενους εδώ πέρα. Και και η κυρία Ματσόνη βεβαίως ήταν παρούσα. Είχαμε λοιπόν συνάντηση με τις αρχές και θέλω να τονίσω πως και ο Υπουργός της Περιφέρειας, ο Ρωμάνο, και ο νέος δήμαρχος της Νάπολης, ο Ντεμάτζιστρης, μας είπαν πως αναμένουν τώρα βελτιώσεις. και πρέπει να επενέσουμε την Άπολη για αυτά τα οποία έκανε σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Τώρα μαζεύουν σκουπίδια πόρτα-πόρτα, προσπαθούν να τα επεξεργαστούν και δεν έχουν απλά χτίσει ε, ένα εργοστάσιο αποτέφρωσης που αργότερα θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά δεδομένου του ότι έχουν περάσει μόνο δύο χρόνια, πρέπει, νομίζω, να επενέσουμε αυτή την πρωτοβουλία και τουλάχιστον ο υπουργό Ρωμάνο θεωρεί πως κομματικές συγκρούσεις δεν πρέπει να καταστρέψουν ε, την υπόθεση αυτή. Δηλαδή, στο παρελθόν θεωρούσαμε πως η χιτά είναι το μέλλον, αλλά η χιτά προκάλεσαν προβλήματα στην καμπανία. Ζητήματα που δεν έχουν λυθεί. Λυπάμαι που δεν ήρθε ο Πίτερ Γιάννα αυτή τη φορά. Γιατί νομίζω πως ε, θα ήταν ενδιαφέρον το ταξίδι. Αλλά επιλογή του ήταν να μην έρθει. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να σας παρουσιάσουμε την έκθεση τον Δεκέμβριο και ευχαριστώ και τη γραμματεία ε, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Και κάτι άλλο πρέπει να συμπεριλάβουμε είναι η πρώτη φορά που έχω πάει σε ταξίδι με ταυτόχρονη διερμηνία και ήταν κάτι το εξαιρετικό αυτό. Ήμασταν πάρα πολύ πιο αποτελεσματικοί με την ταυτόχρονη διερμηνία γιατί σήμαινε πως ε, και το προσωπικό μας επίσης ε, μπορούσε να, να λάβει μέρος. Ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά τα πράγματα λοιπόν με την ε, ταυτόχρονη διερμηνία και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Ε, εντάξει, κάποιο πρέπει να κουβαλάει τον εξοπλισμό, αλλά γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο και είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολτιέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο την κυρία ε, που μας παρουσίασε ορισμένες ε, πτυχές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες από αυτή την επίσκεψη στην Ιταλία. Κάποιοι ε, βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε εκείνη την περιφέρεια έλαβαν μέρος. Θέλω να διευκρινίσω δύο σημεία που αναδύθηκαν από την επίσκεψη, κατά την απόψή μου και πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και στην τελική έκθεση. Καταρχήν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς, όπως είπε και συνάδελφος, βρισκόμαστε ενώπιον μιας σκανδαλώδου έλλειψης ανάληψης ευθύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση που ουσιαστικά δεν ε, σέβονται καθόλου τα πρότυπα της ε, ε, διαλογής και της ε, του διαχωρισμού των αποβλήτων. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα και μάλιστα ακόμη και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος ε, ανακοίνωσε ότι πρέπει να δοθεί κάποια όθηση στην ανάπτυξη αυτού του ζητήματος. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που ανέκυψε κατά την άποψή του και αφορά το μεγαλύτερο μέρος ε, των αναφορών που έχουμε για αυτή την περιοχή. Ποια μεταβατική λύση είναι η πλέον κατάλληλη προκειμένου να επιταχύνει ε, την μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο καθεστώς συλλογής ε, των αποβλήτων. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ο τοπικός επίτροπος, ο οποίος ε, έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτής της μετάβασης ε, έχει εξεύρει μία λύση που κατά τη δική μας άποψη αλλά και την άποψη των αφαιρώτων πηγαίνει ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή δεν διευκολύνει το αντίθετο παρουσιάζει κάποια εμπόδια στο να φτάσουμε σε μία ευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο δηλαδή η λύση να υπάρχει ε, μία χωματερή 18 μηνών που θα διαρκέσει 18 μήνες ε, και θα είναι προσωρινή, τελικά αυτό δεν βοηθά. Έτσι λοιπόν η δράση αυτού του Επιτρόπου ήταν εντελώς μη ικανοποιητική γιατί αυτή η μεταβατική χωματερή θα γίνει μία ακόμη νιωστή οριστική χωματερή και τελικά ε, δεν θα μπορέσει ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση να φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχωρισμού των αποβλήτων. Επομένως, ήδη βλέπουμε ότι έχουμε μία διέξοδο για να αποφύγουν οι αρχές να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επομένως, εδώ βλέπουμε ότι το πραγματικό αδύναμο σημείο και ε, από την πλευρά του Επιτρόπου αλλά και από την πλευρά του Υπουργού εγώ νομίζω δεν έχει αναλυφθεί επαρκής ε, δράση ούτε από τον ε, Υπουργό Περιβάλλοντος. Πρέπει να τονιστεί λοιπόν αυτό το θέμα στη δική μας έκθεση. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω μόλις ε, είχαμε μία νέα πρόταση ε, που θα επιθυμούσαν και οι αναφέροντες ε, και να υπάρχει δυνατότητα όχι μόνο καταγγελίας του προβλήματος αλλά και παρουσίασης εναλλακτικών λύσεων. Πέρα από αυτήν την δημιουργία της χωματερής μεταβατικού χαρακτήρα όπου θα εναποτεθούν 400.000 τόνοι αποβλήτων. Χάρη στο εξαιρετικό έργο και της δικής μας Επιτροπής που επισκέφθηκε την Ιταλία, έχει προταθεί μία λύση η οποία λέει ότι αν χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ε, χώρων υγειονομική ταφής που υπάρχουν στην περιοχή του Λάτσιο είναι δυνατόν να αποφύγουμε την κατασκευή αυτή τη χωματερή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και η Επιτροπή ε, πρέπει να ε, αποκτήσει το έγγραφο αυτό που εκπώνησαν οι πολίτες και οι αναφέροντες και θα πρέπει να στηθεί και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και στον αρμόδιο Επίτροπο για τη Διαχείριση ε, των αποβλήτων στην περιοχή. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μιλάνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά να προσθέσω. Και εγώ παρακολούθησα το έργο της Επιτροπής. Η συνάδελφος ε, Άουκεν ε, πολύ καλά παρουσίασε πώς έχουν τα πράγματα. Ακόμη και αν αυτό το κλίμα της σύγχυσης σε θεσμικό επίπεδο μας οδηγεί στο να αναθέσουμε κάποιες ευθύνες. Μπορώ να σας πω ότι το ζήτημα κυρίως επικεντρώνεται στον ε, αρμόδιο αυτό επίτροπο για την ε, διαχείριση των αποβλήτων. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό ζήτημα, γιατί όπως είπε και ο κ. Γκουαλτιέρη, αυτός ε, ο Επίτροπος απλώς προσπάθησε να δημιουργήσει μια νέα χωματερή, ένα νέο χώρο υγειονομικής ταφής. Τίποτα δεν έκανε για ε, την... Ε, για το διαχωρισμό των αποβλήτων ε, και εμείς επισκεφθήκαμε και την εγκατάσταση του ΆΜΑΚ που δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε αλλά και την εγκατάσταση της Μαλαγκρότα που σήμερα χρησιμοποιείται στο 20% των δυνατοτήτων τους. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτό το φάκελο στην υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ανοιχτή λοιπόν η φάκελη και πρέπει να διατηρηθεί η έκθεση η, αυτή, η αναφορά αυτή η ανοιχτή και νομίζω ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε αν τελικά ε, πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία επί Εγώ νομίζω, και το λέω σιταλός, Ιταλός, ότι θα πρέπει να παραμείνει η διαδικασία επιπαραβάση σε ό,τι αφορά τη χρήση της ε, χωματερής, ε, όπου εκεί εναποτίθεται απόβλητα που δεν έχουν διαχωριστεί, δεν έχουν γίνει αντικείμενο διαχωρισμού. Αν ε, θα ακολουθηθεί ως επιλογή του Μόντι Τελοτάτσο που αναφέρει και ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη αυτό θα πρέπει να γίνει ε, υπό ορισμένε επιφυλάξεις. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι λένε και οι τοπικές αρχές και αν αυτή η επιλογή συνεχίσει να υφίσταται, εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει η ίδια να ε, απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη σπίτι πρέπει να γίνει για αυτή τη διαδικασία παραβάση. Η οδηγία σχετικά με τα πόβλητα είναι σαφής. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση αυτή και διαβούλευση με τους πολίτες πέρα από τα επιστημονικά στοιχεία και τα τεχνικά στοιχεία που μπορούμε να έχουμε αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει να γίνει αυτή η ιδέα της διαχείρισης μέσω επιτρόπου ουσιαστικά είναι σαν να επιβάλλεται ένας ε, αυτοκράτορας, ε, να σκεφτόμαστε ότι ένας ε, επίτροπος μπορεί να παρακάμψει οποιοδήποτε είδος νομοθεσίας. Ένας επίτροπος πρέπει να σέβεται την νομοθεσία για να επιταχύνει τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ο φάκελος πέρα από την έκθεση που θα υλοποιήσουμε και που θα αποσταλεί, και να περιμένουμε, να διατηρήσουμε αυτό το φάκελο ανοιχτό χωρίς να περιμένουμε την επόμενη αναφορά. Αυτό και σε ό,τι αφορά και τη Ρώμη, συγκεκριμένα πολύ, αλλά και το πιο πολύπλοκο θέμα που αφορά ολόκληρη την επικράτεια, ολόκληρη την επαρχία. Και να κλείσω εν συντομία. Όταν ε, εμφανίζονται τέτοιες ε, συμπεριφορές παντοδυναμίας, τότε η στάση αυτού του επιτρόπου θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κατασκευαστεί γενιωστή φορά φορά ε, μια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού για να απαντήσουμε στις ανάγκες της Ρώμης. Όμω, ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα, ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται στις δυνατό, στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Και δεν γίνεται τίποτα για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι εγκαταστάσει εκείνε και σκεφτόνται να κατασκευάσουν κάτι καινούριο. Μια νέα εγκατάσταση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Γιατί και σε αυτό το θέμα η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει ειδική αναφορά, συγκεκριμένη αναφορά και οι αναφέροντες τη δεύτερη μέρα της συνάντησής μας μας δήλωσαν ε, την ανησυχία τους γιατί σε εκείνη την περιοχή Υπάρχουν, ε, είναι ήδη η περιοχή αυτή βεβαρημένη ε, με βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν ε, και χημικές βιομηχανίες που έχουν μολύνει πάρα πολύ τα υπογεΐδατα. Και έχουμε και παρουσία χωματερής και έχουμε και παρουσία εγκατάστασης αποτέφρωσης των αποβλήτων. Επομένω, ε, αν είχαμε μια αναγκατάσταση θα ζημιωνόταν περαιτέρω αυτή η περιοχή. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να καταρτήσουμε μια πάρα πολύ αυστηρή έκθεση κατά των συμπεριφορών αυτών, κατά των δράσεων αυτών ε, και ε, εντάξει συμφωνώ με οσοι υπόθηκαν από την κυρία Όκεν ότι υπάρχει μια σύγχυση και σε επίπεδο θεσμών. Ο, υπάρχει η ευθύνη τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και του επιτρόπου που έχει διοριστεί αρμόδιο για τα απόβλητα. Θα πρέπει να παραμείνει λοιπόν ο φάκελο ανοιχτό για να δούμε αν οι διάφορε ενέργειε και συμπεριφορέ αυτού του επιτρόπου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασία επί παραβάση. Όχι μόνο για το θέμα τη χωματερή, αλλά και να δούμε αν δεν έχει γίνει σεβαστή η οδηγία για το περιβάλλον και η οδηγία για τα απόβλητα. Τώρα δίνω τον λόγο ε, κυρία Τζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους Γκουαλτιέρη και Μιλάνα. Υπογραμμίζω πολύ σύντομα ότι οι εργασίες μας θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτή την προβληματική του προσωρινού χαρακτήρα χαρακτήρα ε, της τοποθεσίας του Μόρτιν Τελορτάτσο, γιατί η δική μας ανησυχία, αλλά και η ανησυχία των πολιτών, είναι αυτός ο προσωρινός χαρακτήρας, όμως μήπως ε, αντί να παραμείνει προσωρινή ε, αυτή η χωματερή, ουσιαστικά μετατραπεί σε μόνιμη. Και εμείς εναντιονόμαστε κάθετα σε αυτό. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε επίσης ε, το πρόβλημα της ε, προσέγγισης ε, ως κατεπίγουσας κατάστασης. Όπως είπε και ο κύριος Μιλάνα, δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση με τους πολίτες. Επομένως, όλοι οι πολίτες, οι τοπικές αρχές ακόμη και αν εξέφρασαν αρνητική αντίθετη άποψη, και αναφέροντας και συγκεκριμένη τεκμηρίωση και μέσω συλλογής υπογραφών, δεν ακούστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ε, στις ε, αρχές που έπρεπε να λάβουν την απόφαση τη σχετική τεκμηρίωση, τα σχετικά έγγραφα, τα αποδεικτικά που είχαν συλλέξει. Απλώς ε, μία διαβούλευση έγινε όταν την περασμένη εβδομάδα πήγαμε εμείς ως Επιτροπή Αναφορών στην Ιταλία. Αυτό μεταξύ άλλων έρχεται σε αντίθεση και με τις προσδοκίες ε, του τοπικού πληθυσμού που στο κλείσιμο της ε, Μαλαγκρότα έβλεπαν ότι τελικά θα δινόταν τέλος ε, στην ε, περιβαλλοντική λαϊλασία ε, αυτής της τοποθεσίας. Οι πολίτες περίμεναν ότι με το κλείσιμο της Μαλαγκρότα τελικά θα ξεκινούσε μια στρατηγική αποκατάσταση όλης της περιοχής της Κοιλάδας Γαλέρια, αλλά Τελικά, αν κλείσει η Μαλαγκρότα και ανοίξει το Μόντι Ντελορτέτσο με ένα προσωρινό χαρακτήρα 18 μηνών, τι να σα πω, το θέμα είναι ότι κανεί δεν πιστεύει σε αυτόν τον προσωρινό χαρακτήρα. Επομένως, Θέλω να συγχαρώ όλη την Επιτροπή Αναφορών, γιατί εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους ε, παρακολουθήσαμε ε, τις ε, εργασίες, γιατί δεν είμαστε τακτικά μέλη, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάνετε μια δουλειά που την εκτιμά πάρα πολύ ο κόσμος, οι πολίτες και εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει η Επιτροπή Αναφορών αλλά και γενικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. No, σας ευχαριστούμε κυρία Αντζελίνη. Δίνω τώρα τον λόγο στον κύριο Μπουστινάρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτη διαπίστωση. Η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών να αποστείλει ε, μια νέα αποστολή ε, για ενημέρωση στην Ιταλία υπήρξε μια πάρα πολύ καλή απόφαση. Πρόκειται για μια απόφαση που βασίστηκε σε μια εξέλιξη η οποία παραμένει ανησυχητική στην Ιταλία. Επιπλέον, τις ε, λάβαμε σήμερα πληροφορίες σημαντικές που επιβεβαιώνουν ότι η απόφαση αυτή ήταν πάρα πολύ εύστοχη, είναι πολύ έντιμη προσέγγιση, είναι δίκαιη και όσοι ε, συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη τη συμμερίζονται, είτε πρόκειται για μέλη ε, της ομάδας ε, που επισκέφθηκε την περιοχή αυτή, είτε πρόκειται για τους Ιταλούς συναδέλφους. Είναι λοιπόν μια επιτυχία, κυρίως επειδή πρόκειται για ένα θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο τεταμένων συζητήσεων στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, θα ήθελα να επιμείνω πάνω στην σοβαρότητα, στην μεγάλη σοβαρότητα της περίπτωσης αυτής. Ας μην ξεχνούμε ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά ένα έδαφος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για ένα κράτος μέλος, ένα ιδρυτικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το κράτος άλλη μια φορά η διερευνητική αποστολή διαπίστωσε όχι μόνο την μη συμμόρφωση αλλά και την συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας και της εθνικής και της ευρωπαϊκής που αφορά το θέμα που μας απασχολεί. Και αυτό βεβαίως ανησυχεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά αυτό θα πρέπει επίσης in να καταλήξει σε μια αντίδραση των αρμοδίων αρχών για να μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα. Τρίτον, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν λαμβάνει χώρα σε μια χώρα που έχει μειωμένη ικανότητα διοικητική και τεχνολογική. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα κράτη-μέλη, από τα πλούσια κράτη-μέλη, από τα κράτη που έχει μεγάλη ικανότητα τεχνολογική, βιομηχανική μεγάλες δυνατότητες. Εξού και η μεγαλύτερη ανησυχία μου, εξού και η οδύνη μου, διότι είμαι μεγάλος φίλος της Ιταλίας, εξού και το σοκ που αισθάνομαι βλέποντας αυτή την πραγματικότητα. Έχω την εντύπωση ότι ίσως έρχεται, είναι εικόνες ε, του φιλμ Shocking Asia, ίσως ακούσατε την ταινία αυτή. Αυτά συμβαίνουν το 2012 σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Τέταρτον, θα ήθελα ειλικρινά να πω ότι χαίρομαι για την συμβολή όλων των συμμετεχόντων μονίμων μελών αλλά και ε, αναπληρωτών διότι μαζί συνέταξαν μια καλή δίκαιη ισορροπημένη έκθεση που ε, τονίζει τις δυνατές λύσεις ε, για να βγούμε από αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει με αυστηρότητα να εντοπίσει τις ευθύνες, ένα πρόγραμμα δράσης και τις προθεσμίες που θα πρέπει να επιβληθούν σε συνεργασία με τις τοπικές περιφερειακές και εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συμβάλλει στο να δοθεί τέλος σε αυτήν την τελείως απαράδεκτη κατάσταση. Και τέλος, και αυτό είναι σημαντικό, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο αντικείμενο που με ανησυχεί αυτού του είδους της διαχείρισης εντός εισαγωγικών του προβλήματος των αποβλήτων τίνει να εξάγεται. Και μπορώ αυτή τη φορά να σας πω ότι οι πληροφορίες που παρουσίασε ο τύπος στη Ρουμανία επιβεβαιώνουν ότι Ιταλικά απόβλητα εξάγονται και ο, ο τύπος στην Ρουμανία μας λέει ότι πολύ συχνά ε, μέλη της Ιταλικής Μαφίας εμπλέκονται σε αυτές τις μεταφορές και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την Επιτροπή κατά του οργανωμένου εγκλήματος να ζητήσω από όλα αυτά τα όργανα να παρακολουθήσουν εκ του σύναγγης το θέμα αυτό με πάρα πολύ σοβαρότητα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται ένα τέτοιο μοντέλο, ένα τέτοιο μοντέλο που να οδηγεί στην πτώχευση, ένα τέτοιο καταστροφικό μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων που εξυπηρετεί το συμφέρον μερικών και που είναι καταστροφικό για όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα δίνω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και μετά στην κυρία Όκεν για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει τον λόγο. Κύριε Κοντέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί πάρα πολύ για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων στην Ιταλία και για τον λόγο αυτό. Ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση ε, κατά της Ιταλίας ε, και ήδη προετοιμάζονται και κάποιοι Σχετική φάκελη. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές, ειδικά στο κεντρικό επίπεδο, αλλά όπως ε, σωστά ευσημάνθηκε υπάρχουν ε, πολλές αρμοδιότητες και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και μέρος του προβλήματος είναι ε, αυτό που αφορά την εφαρμογή. Για το θέμα τώρα των παράνομων χωματερών Όπω ξέρετε η υπόθεση αυτή έχει προχωρήσει πολύ. Η Κομισιόν αποφάσισε να προσφύγει δεύτερη φορά στο δικαστήριο ζητώντα πρόστιμα. Αυτό είναι. Η υπόθεση είναι πολύ παλιά. Έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχει η Κομισιόν, έχει μειωθεί ο αριθμό των παράνομων χωματερών, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ εκτεταμένο το πρόβλημα ε, και αφορά πολλέ περιφέρειες στην Ιταλία. Ε, εξού και η κίνηση αυτή της Κομισιόν. Υπάρχει άλλη μία παράβαση εδώ και καιρό που αφορά την καμπανία. Υπάρχει απόφαση του ΔΕΚ ε, πριν από δύο χρόνια. Το δικαστήριο θεώρησε πως η Ιταλία έχει παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο, την οδηγία πλαίσιο και επίσης απειλείται και η υγεία των κατοίκων της περιοχής και το περιβάλλον. Οπότε παρακολουθούμε στενά την κατάσταση είχαμε κάποια πρόοδο. Αυτό το οποίο εξετάζουμε τώρα είναι το εάν η πρόοδος αυτή είναι επαρκής και αν η απειλή προς την υγεία είναι ελεγχόμενη βραχυπρόθεσμα και μέσω πρόθεσμα θα υπάρξει βεβαίως ένα δίκτυο διαχείρισης ε, των αποβλήτων της καμπανίας. Για το ζήτημα της Μαλαγκρότα, όπως ξέρετε, η Κομισιόν έστειλε μια αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία τον Ιούνιο για την έλλειψη επαρκούς προ επεξεργασίας των αποβλήτων, γιατί ξέρετε πως το ζήτημα αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την ε, Μαλαγκρότα. Τον Αύγουστο λάβαμε την ε, απάντηση των Ιταλικών αρχών, την αξιολογούμε και τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από αυτό. Αλλά ανησυχούμε και για το ζήτημα της ε, Μαλαγκρότα και, και παραπέρα γιατί όπως είπαμε ε, ο τεράστιος αυτός χιτά έχει φτάσει στο τέλος του χρόνου ζωής ε, και ενδιαφερόμαστε για το τι θα γίνει με την επόμενη λύση για την διάθεση των αποβλήτων. Αυτό το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι πως ε, οι λύσεις και τα σημεία στα οποία θα εφαρμοστούν δεν ε, είναι δουλειά της Κομισιόν, δηλαδή το ποια θα είναι η λύση και το πού θα εφαρμοστεί, αρκεί να ε, συμμορφώνεται με την ε, νομοθεσία. Ε, είμαστε σε επαφή με τις Ιταλικές Αρχές και επισημάναμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη, η λύση που θα ακολουθήσει την Μαλαγκρότα να εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δικαίο. Παραδείγματος χάρη να γίνει δικαιο του χαρη αξιολόγηση αντικτύπου, και δημόσια διαβούλευση. Επίσης παρακολουθούμε και το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων στο Λάτσιο γιατί η Ιταλία υιοθέτησε ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων οπότε τα εργαλεία υπάρχουν τώρα πρέπει να, να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο Οπότε να πω πως η Κομισιόν ενδιαφέρεται για την πρόοδο αυτών των ζητημάτων και δεν θα διστάσει να κάνει τα αναγκαία βήματα εάν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω και εγώ κάτι αλλά παρακαλώ σύντομα όποιο θέλει να μιλήσει γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει και η συνεδρίαση των συντονιστών. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ιταλούς συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ήταν χρήσιμο το ότι ήταν ε, παρόντες ε, στην επίσκεψη και αποφασίσαμε πως η επίσημη αντιπροσωπεία βεβαίως δεν θα πρέπει να αποτελείται από βουλευτές ε, από την εν λόγω χώρα γιατί έτσι έχουμε και μεγαλύτερη αξιοπιστία γιατί ο κόσμος το βλέπει και κομματικά οπότε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ως κάποιος εξωτερικός, αντικειμενικός παρατηρητής ε, ο κόσμος αισθάνεται πως υπάρχει σωστή ε, μεταχείριση και όταν κάνουμε αυτό που κάναμε στην Ιταλία όπου οι Ιταλοί συνάλφοι ήταν ε, παρόντες ε, και στις ε, συναντήσεις στη Ρώμη. Νομίζω πως ήταν αρκετά καλό το μήνυμα και για τις μελλοντικές μας αποστολές. Και κάποια πιο συγκεκριμένα τώρα σχόλια. έχει σημασία εδώ πέρα η στρατηγική της Ιταλίας. Δηλαδή όταν συσσωρευτούν τα σκουπίδια λένε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ε, και παραμερίζουν όλη την νομοθεσία και τα πετάνε στην κοντινότερη χωματερή που συνήθως είναι και μια πολύ ωραία περιοχή αλλά ε, δεν θα παραπονεθούν οι άνθρωποι ξέρω εγώ ή δεν θα θυχτούν οικονομικά συμφέροντα πρέπει να το δούμε αυτό δηλαδή αυτή η έννοια της εκτάκτου ανάγκης ε, πρέπει να τελειώσει και αυτή δεν είναι δυνατόν δεν μπορούμε να παραμερίζουμε και την ομοθεσία φωνάζοντας ε, κατάσταση ανάγκης και κάτι ακόμα. Το ένα είναι αυτό το οποίο επεσήμανε ο Βίκτορ για την εξαγωγή των αποβλήτων. Είναι σαφές ε, πως ε, υπάρχουν ακόμα μαφιόζικα συμφέροντα στις μεταφορές και δυστυχώς αν το ερευνούσαμε παραπέρα θα βλέπαμε πως ε, οι βιομηχανίες της Βόρειας ε, Ιταλίας ε, χρησιμοποιούν τη μαφία για να ξεφορτωθούν τα απόλυτα αντί να πληρώσουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτό το οποίο γίνεται τώρα στην Άπολη είναι πως κάποια σκουπίδια στέλνονται για αποτέφρωση στην Ολλανδία και ίσως να είναι έξυπνη αυτή η στρατηγική. Αντί δηλαδή να αυξάνεται, να αυξάνεται υπάρξουν εγκαταστάσεις ε, ε, αποτέφρωσης στην Νάπολη πρέπει να χρησιμοποιήσουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οδηγία των αποβλήτων για να αυξηθεί η ανάκτηση, η ανακύκλωση κτλ. Και νομίζω μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως το πρόβλημα είναι σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Δανία θα συμφέρει να, να αποτεφρώνουμε τα πάντα οι πυρομανείς εκεί πέρα της Βόρειας Ευρώπης. Και η στρατηγική μας αυτή, δηλαδή της αποτέφρωσης για παραγωγή ενέργειας, ε, έχει υποκαταστήσει κάτι άλλο. Οπότε δεν πρέπει να κοιτάμε την Ιταλία ε, μόνο για μαφία, αλλά να κοιτάξουμε λίγο και τη Βόρεια Ευρώπη και κάποιε δραστηριότητε που κάνουν. Και η Τζούντιθ Μέρκη δεν ήταν υπέρ τη αποτέφρωση. Τέλο, ε, για τα λεφτά, όποτε, ζητάμε, όποτε συναντιόμαστε με του Ιταλού, ε, ζητάνε λεφτά και Κομισιόν. Είπε πρέπει να δούμε πρώτα αξιόπιστα σχέδια. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία είδαμε είναι απλά φαντασία. Είδαμε όμως κάτι το οποίο ήταν απτό στην Άπολη, δεν ήταν φαντασία και μου είπαν και κάτι άλλο εκεί πέρα από την περιφέρεια και παρά το ότι γνωρίζω βεβαίω πως είναι δουλειά της Ιταλίας να μοιράσει τα λεφτά ε, νομίζω πως πρέπει να γράψουμε στην έκθεση πως τις ε, περιοχές όπου γίνονται θετικά βήματα καλό είναι να τις στηρίζουμε οικονομικά για να εφαρμόσουν τα θετικά αυτά σχέδια. Θέλω να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεση. Γιατί βλέπουμε πραγματική πρόοδο. Ευχαριστώ. Κύριε Μιλάνα, σας παρακαλώ να είστε και εσείς πάρα πολύ σύντομος. Μόνο μια ερώτηση στην Κομισιόν. Τον Ιούλιο είχαμε μια άλλη ακρόαση για μια άλλη περίπτωση για το Κορκόλε, πάντοτε στην περιοχή του Λάτσιο και η Κομισιόν μας υποσχέθηκε να παραγγείλει από την Επιτροπή Αναφορών μία έκθεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε ποιο σημείο βρίσκεται η έκθεση αυτή, γιατί πρέπει να πούμε ότι το Λάτσιο είναι υποπαρατήρηση, υποπαρακολούθηση, εμείς περιμένουμε τι απαντήσει του Αυγούστου και αμέσω μετά θα έχουμε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην Επιτροπή ΠΕΤΗ. Εγώ θα ήθελα να σταλεί η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να σταλεί και κάτι ακόμη. Πώς έκλεισε η διαδικασία επί παραβάση για το Λάτσιο. Δηλαδή, αν το σχέδιο για το οποίο συζητάμε ή ε, πραγματικά το αμφισβητούν τόσο πολύ και το ακούσαμε σήμερα το πρωί. Προβλέπετε μία νέα χωματερή στο Μοντετελετάτσο. Προβλέπετε στο σχέδιο αυτό να υπάρχει βιολογική ε, επεξεργασία ε, των αποβλήτων και υπάρχουν όμως όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε εμείς εντοπίσει σήμερα για τη μαλαγκρότα. Και ρωτάω, αυτό το σχέδιο ποια αξιοπιστία είχε αν σήμερα οι πολίτες ε, και η Επιτροπή Αναφορών που το υπολήθευσε, αν ε, οι θεσμοί καταγγέλουν ένα τέτοιο σχέδιο, μήπως θα έπρεπε ε, να δούμε εδώ ποια είναι η στάση της Κομισιόν απέναντι στη χώρα αυτή, μήπως δεν είναι τόσο κάθετη όπως θα έπρεπε. Η κυρία Τζελίλη. Και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση πάντοτε στην Κομισιόν. Θεωρώ ότι η Κομισιόν για νιωστή φορά θα έπρεπε να πει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή θέλει να εγγυηθεί στους πολίτες τη δυνατότητα πραγματικά να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ακόμη και αν ε, τελικά επιλεγεί αυτή η τοποθεσία, βλέπουμε όμως ότι μέσα στη διαδικασία προς το παρόν έχει υπάρξει άρνηση του δικαιώματος ε, των πολιτών να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε δύο λεπτά διάλειμμα για να περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών που θα λάβει χώρα και κλεισμένων των θυρών